Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Θυμίζω ότι το πρώτο μέρος της ήταν και κλεισμένο των θυρών για να ακούσουμε κάποιες μαρτυρίες και θεώρησαν οι ενδιαφερόμενοι ότι ήταν καλύτερο να είναι και κλεισμένο των θυρών. Τώρα έχουμε μια μισή ώρα συζήτηση με κάποιους εκπροσώπους του Διεθνούς Κονσόρσιου Δημοσιογράφων που ε, ασχολούνται με την ερευνητική δημοσιογραφία. Ζητάει το λόγο ο κύριος Μάζη, Φάμπιο. Θα ήθελα κάτι να διορθώσω. Μια ενημέρωση, μια πληροφορία που δώσατε. Η Γαλλίδα καταγγέλουσα μόλις μας είπε ότι θα ήθελε να κάνει δήλωση δημόσια. Οπότε έγινε κάποια παρεξήγηση μάλλον. Και θα ήθελα αυτό να διευκρινιστεί. Ο πρόεδρος. Ωραία. Θα διευκρινιστεί, αγαπητέ Φάμπιο. Είχε συμφωνηθεί με τη γραμματεία και τους ενδιαφερομένους και προέβλεπαν κατόπιν δικού τους αιτήματο να είναι και κλεισμένο το θυρώνη συνεδρίαση. Εγώ ο ίδιος ερχόμενος ρώτησα και τους δύο. Οπότε ο καθένας ε, είναι ελεύθερος να αλλάξει γνώμη και εδώ στην κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίαση. Μετά τη συνεδρίαση είχαν την ευκαιρία οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επαφή με όλους τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες και να κάνουν τα δημόσια σχόλια που θεωρούσαν σκόπιμα. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω για να κάνουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Λοιπόν, επειδή διεπόμεθα από ε, αυτή την ε, έγνοια για διαφάνεια, καλωσορίζω σε δημόσια συνεδρίαση τους δημοσιογράφους, η οποία δημόσια συνεδρίαση μεταδίδεται και απευθεία στο διαδίκτυο ε, από την ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και το δικό μας ιστότοπο της ε, ειδική ε, Προσωρινής Επιτροπής. Έχουμε τους δημοσιογράφους που είναι οι εξή κύριοι. Κρίστοφ Κλέριξ, Εντουάρ Περά, Ρίτσαρτ Μπρούξ, Λάξ Μπουβέ και Ξαβιέ Κουνάς. με την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε προηγουμένως θα ζητήσω από τους δύο εισηγητές μας να κάνουν πρώτα ερωτήσεις και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους ε, κυρίους δημοσιογράφους. Δύο εκπρόσωποι τους θα καταθέσουν τη μαρτυρία τους και μετά θα ξαναδώσω ε, το λόγο σε έναν εκπρόσωπο κάθε πολιτικής ομάδας. Όσο γίνεται πιο σύντομα για να ε, έχουμε ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση. Να αρχίσουμε τώρα από την Ελίζα γιατί προηγουμένω μίλησε πρώτος ο Μίχαελ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας κατευχαριστήσω που είστε εδώ ε, είναι πολύ χρήσιμο να ακούσουμε τις συνεισφορά σας και ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε στα χέρια μας τα απορίσματα της δουλειάς σας. Συγχαρητήρια που υπήρξατε θαραλέοι και κάνατε αυτές τις αποκαλύψεις. Τώρα πιο συγκεκριμένα αυτό που ήθελα να μου πείτε είναι εάν έχετε δημοσιεύσει τις περισσότερες πληροφορίες που λάβατε και αν σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτό το είδος δουλειά. τι όθηση να δώσουμε εμείς για να μπορέσετε να αναπτύξετε περισσότερο όσο έχετε ήδη κάνει. Στην Ευρώπη ασχολούμαστε με θέματα που μπορεί να είναι ε, νόμιμα ή ανήθικα και ε, παράνομες πρακτικές. Πώς το βλέπετε αυτό από πολιτικής σκοπιάς προσπαθούμε να ε, προσεγγίσουμε το πολιτικό ε, ηθικών με το νόμιμο. Όμως εδώ υπάρχουν κάποιες πρακτικές που είναι στα όρια της παρανομίας και που μας βοηθήσατε κι εσείς να τις κατανοήσουμε. Πώς βλέπετε τη φορολογία στην Ευρώπη επίσης. Υπάρχουν συνήθεις ύποπτοι όπως θα μπορούσαμε να τους πούμε, αλλά έχετε περισσότερες πληροφορίες για την όλη κατάσταση στην Ευρώπη περιφορολογικών. Τι γίνεται με τις ε, εταιρείε offshore επίσης, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα με σοβαρότητα. Και επίσης ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προτάσεις σας για τη δική μας τη δουλειά. Τι γίνεται με τις εταιρείε λοιπόν της υπεράκτης η όλη συζήτηση αυτή θα μπορούσε να συνεχιστεί. Ε, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές συστάσεις για ποτέ βρείτε το θέμα της ε, φορολογίας. Τι προτείνετε για τη μελλοντική μας δουλειά λοιπόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να σας έχουμε στο πλευρό μας ως ε, εταίρους και συνομιλητές στην διαδικασία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Τόιρερ. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρώτα θα ήθελα να επισημάνω ότι μόλις πριν λίγο στεκόμουν δίπλα στην καταγγέλουσα κυρία Ζιμπό όταν ήταν και ο κύριος Διμπάζη ε, κοντά της και η ίδια πράγματι είπε ότι ήταν διατεθειμένη να κάνει και δημόσια δήλωση. Αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Απευθύνω το καλώς ορίσατε στους εκπροσώπους που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι μέσω της θαραλέας δημοσιογραφικής στάσης τους απεκάλυψαν πράγματα τα οποία πολλοί δεν μπορούσαν να τα φανταστούν. Είναι λοιπόν προφανές ότι γίνονται, υπάρχουν επιθετικά μοντέλα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στα οποία βασίζονται και έτσι πετυχαίνουν σημαντικότατες μειώσεις των φορολογικών βαρών τους μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και όμιλοι. Στην, ε, σε αυτό το πλαίσιο μας ενδιαφέρει να μάθουμε εάν κατά την ανάγνωση των εγγράφων που έχετε κάνει περιλαμβάνονται και κάποιες παραπομπές στο έργο των νομοθετών που μέχρι τώρα δεν μπορέσατε να αξιολογήσετε. Ε, κάνατε τον κόπο εσείς οι ίδιοι να αναλύσετε ορισμένες χιλιάδες σελίδων Ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές ε, τις ε, χρησιμοποίησατε και δημοσιογραφικά. Εμείς θέλουμε να μάθουμε ποια από τα πράγματα αυτά ήταν νόμιμα, ποια ήταν τα παράνομα και πού ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα. Εδώ βεβαίως τίθεται και το θέμα του ρόλου των χωρών μελών. Δεν είναι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα όργανα εκείνα που δήθεν εμπόδισαν τις χώρες μέλη να συνεργαστούν καλύτερα στην διερεύνηση των φορολογικών υποθέσεων. Οι χώρες μέλη είναι εκείνες οι οποίες παραλείπουν εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Γι' αυτό η ερώτησή μου προς εσάς, πού θα πρέπει να αρχίσει ο νομοθέτης. Πώς κρίνεται επίσης τον ρόλο των τεσσάρων μεγάλων φορολογικών συμβούλων εννοείται και πώς κρίνεται τον ρόλο των ενδιαφερομένων χωρών. Τέλος, ο ρόλος των καταγγελόντων, ο ρόλος των προστατευόμενων μαρτύρων. Μόλις πριν μάθαμε από δύο από τους μάρτυρες αυτούς ποια ήταν η μοίρα των καταγγελόντων αυτών μετά από την καταγγελία των παράνομων πράξεων στην οποία προέβησαν. Και τι, πώς κρίνεται την ποινική διοξή τους. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος προβαίνει σε καταγγελίες σε μια χώρα μέλος για φόρο διαφυγή, να διώκεται ποινικά σε άλλη χώρα μέλος. Αυτό είναι αντίθετο με οποιοδήποτε αίσθημα δικαιοσύνης. Γι' αυτό και ρωτώ, απευθύνω ερώτημα προς εσάς, τι πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη σας μέσα από τις εμπειρίες σας έτσι ώστε να προστατευτούν καλύτερα οι καταγγέλλοντες και έτσι ώστε να γίνει και ισχυρότερο το κίνητρο αποκάλυψης παράνομων δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους σας 10 λεπτά για να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση. Ο κύριος Πέγα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Εγώ άρχισα να ερευνώ αυτό το θέμα το 2011 το καλοκαίρι. Όλοι μου οι συνομιλητές τότε ε, μιλούσαν για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, για φορολογική βελτιστοποίηση. Ε, έλεγαν ότι είναι νόμιμο, βέβαια δεν είναι πάρα πολύ ηθικό. Υπήρχαν τέτοια εργαλεία και πολύ γρήγορα εγώ έμαθα για αυτά τα rulings, ε, κάποιες εχέμηθες συμφωνίες φορολογικές μεταξύ εφορίας και εταιριών και πολλές πηγές μου είπανε ότι διακρινότανε το Λουξεμβούργο τότε σε αυτή την προσπάθεια στις επιδόσεις και άρχισα να το ερευνώ. Το Μάιο του 2012, μετά από διάφορες φορολογικές συμφωνίες που ήρθαν στα χέρια μου, δημοσίευσα μια πρώτη έρευνα ε, στο γαλλικό κανάλι ε, France 2 στην τηλεόραση. Ε, είχα πολύ σημαντικά στοιχεία ήδη και συγκεκριμένα έγγραφα που ήταν πάρα πολύ τεχνητά πολλέ φορέ για να πληρώσουν λιγότερους φόρους οι εταιρείε. Για πρώτη φορά αυτά τα rulings λοιπόν έβγαιναν στη δημοσιότητα. Μία μόνο συνέντευξη τύπου έδωσε ο τότε Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου και καμία δεν ήταν στη συνέχεια πολιτική αντίδραση. Πουθενά. Τον Ιούνιο του 2013, μετά από νέα στοιχεία, πάντα στη France 2, στο ίδιο γαλλικό κανάλι, δεύτερη έρευνα, σιγή ηχθείω. Καμία πολιτική αντίδραση ούτε στη Γαλλία ούτε πουθενά στην Ευρώπη. Χρειάστηκε διεκτή έρευνα και τα LuxLeaks το Νοέμβριο 2014 από του συναδέλφου εδώ παρόντε και άλλου που δεν είναι εδώ, για να βγει αυτό το καυτό θέμα, να γίνει δημόσιο και να αποκτήσει τη σημασία που του αξίζει. Η Επιτροπή σας είναι άμεση συνέπεια όλων αυτών και σας είμαι ευγνώμων πάρα πολύ που με καλέσατε με τους συναδέλφους για να ε, δώσουμε τη μαρτυρία μας. Λυπάμαι πάρα πολύ και εγώ όπως και άλλοι που το Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να κάνει μια ουσιαστική ε, εξεταστική ερευνητική επιτροπή με τις εξουσίες και τα μέσα που έχει. Στην αρχή αυτό ήθελαν οι ευρωβουλευτές και νομίζω ότι το αξίζουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες και το απαιτεί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Ε, με κάλεσε αυτή η ειδική επιτροπή πριν από λίγους μήνες να έρθω να σας δώσω τη μαρτυρία μου ως δημοσιογράφος. Στις 23 Απριλίου μου άσκησε ποινική δίωξη το Λουξεμβούργο για τη δουλειά μου σε αυτό το θέμα. Και με, δύο μέρες μετά 28 Υπουργοί Οικονομικών αποφασίζουν ομόφωνα να ανταλλάσσουν rulings. Πρώτη πρώτου του 2016 θα τεθεί σε ίσχυ αυτό και ο Πρέ ε, ο Λουξεμβούργιος υπουργό ε, δήλωσε ότι με μανία θα εργαστεί για να είναι έτοιμη η οδηγία εμπρόθεσμα. Ε, συμπίπτουν όλα αυτά χρονικά με τη δική μου δίωξη. Είμαι υπό μια διαδικασία δικαστική δεν μπορώ να αποφανθώ επί της ουσίας του θέματος που με αφορά. Να απαντήσω στις ερωτήσεις, θέλω να σας προειδοποιήσω, απειλούνται όχι μόνο οι καταγγέλλοντες αλλά και οι δημοσιογράφοι που ρισκάρουν να ασχοληθούν με τέτοιου είδους θέματα. Είναι ε, συμπτωματικό και ταυτόχρονα δραματικό ε, να δούμε ότι οι μόνες διαδικασίες και δίκες είναι εις βάρος των καταγγελόντων και όχι εις βάρος των πηγών του προβλήματος ε, και των αιτίων. Ταυτόχρονα σχέδιο οδηγίε για το εμπορικό απόρριτο προετοιμάζεται στι Βρυξέλλε με πολύ ανησυχητικά στοιχεία για το δικαίωμα στην πληροφόρηση των πολιτών για θέματα δημοσίου συμφέροντο και ενδιαφέροντο. Είναι πολύ λίγε οι ασφαλιστικέ δικλείδε για δημοσιογράφου και καταγγέλλοντε. Και το σχέδιο αυτό γινόταν χωρίς καμία διαβούλευση μέχρι πρόσφατα. Για να μας καθησυχάσουν λένε ότι προστατεύονται οι δημοσιογράφοι και οι καταγγέλλοντες όταν αποκαλύπτουν παρανομίες, αλλά στο LuxLeaks δεν είναι παρανομία, γιατί μας λένε αφού είναι όλα νόμιμα. Απλώς ε, βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί οι συμφωνίες του Λουξεμβούργου θεωρούνται νόμιμες αυτά τα rulings. Αυτά ήθελα να σας πω εισαγωγικά. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο φίλο μου Ρίτσαρτ Μπρούξ, ο οποίος με βοήθησε να κατανοήσω αυτά τα περίπλοκα σχήματα του Λουξεμβούργου. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Ευχαριστούμε κύριε Πέρα. Ο κύριος Μπρούξ, ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι ο Ρίτσαρτ Μπρούξ και είμαι δημοσιογράφος του Time, του Eye στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, από το 2012 ερευνώ το θέμα αυτό και δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες του εγγράφου μόνο πολύ σύντομα στοιχεία το βασικό πρόβλημα με το Λουξεμβούργο είναι ότι οι οικονομικές αρχές επέτρεψαν να λειτουργήσει φορολογικός παράδεισος στην καρδιά της Ευρώπης αλλά όχι με την κλασική μορφή του φορολογικού παραδείσου που είναι ένα τροπικό νησί ηλιόλουστο, αλλά ε, ένα κράτος που είναι ουσιαστικά εταίρος των μεγαλύτερων οικονομικών ε, ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΩΣΑ και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίω. Οι πολυεθνικές εταιρείε λοιπόν μπορούσαν χωρίς ε, φορολογικούς να βάζουν και να βγάζουν χρήμα επιφεύγοντα την εφορία της χώρας τους πολλές φορές και με πολύ χαμηλή φορολόγηση στο Λουξεμβούργο. Αυτό θυμίζει πιο πολύ τροπικό φορολογικό παράδεισο, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όμως εμφανώς αλλά και καλυμμένα με τα έγγραφα του LuxLeaks και τις λεπτομέρειες του συστήματος είδατε πως το Λουξεμβούργο προσαρμόζει την χώρια νομοθεσία ώστε να μην φορολογείται το εισόδημα στη χώρα. Έχει βεβαίως 29% εταιρικό φόρο το Λουξεμβούργο, θεωρητικά, είναι αρκετά υψηλός, όμως με τα συγκεκριμένο σύστημα, με αυτές τις συμφωνίες μπορεί να φτάνουν ε, το ποσοστό αυτό στο ένα λεπτό του ευρώ. Με δάνεια υβρίδια, με αλλαγές τομέα εργασιών. Στην ουσία καταλήγουν όλα με τους διάφορους μηχανισμούς του Λουξεμβούργου στο μηδενικό φόρο και όλα έχουν να κάνουν με την ερμηνεία της εγχώριας νομοθεσίας με το γεγονός ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τις λεπτομέρειες των νόμων και ότι είναι πολύ επικής η φορολογική αρχή στο Λουξεμβούργο. Είναι δύσκολο να το αμφισβητήσει κανείς το σύστημα αυτό και ιδιαίτερος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, όπως έχει ανακρίνει κάποιες ε, ήπιες συμφωνίες όπως ονομάζονται, κάποιες ιδιαίτερα βολικές συμφωνίες όπως αυτή της Amazon. Αυτές οι εταιρείες, αρκεί να έχουν ε, το χρήμα που απαιτείται, είναι διαθέσιμες για όλους. Δηλαδή, όσο πιο πολύ χρήμα μπορεί να διαθέσει κανείς, τόσο πιο χαμηλό φορολογικό συντελεστή μπορεί να διαμορφωτευτεί. Αυτό φαίνεται από διάφορα έγγραφα. Δηλαδή, η... τα φορολογικά περιθώρια που δίνει το Λουξεμβούργο είναι... μπορεί να είναι 6 δισεκατομμύρια είναι, αν μπορεί κανείς να δώσει 64 δις, να πάρει ένα 64 του 1% ως φόρο. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν γι' αυτό. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία είναι αυτή του ΩΣΑ και ονομάζεται η πρωτοβουλία για την διάβρωση της φορολογικής βάσης και την αντιμετώπιση της. Είναι μια διαδικασία κάπως βραδικίνητη παρόλο που κάνει την πορεία ΩΣΑ και απαιτεί τα κράτη-μέλη του ΩΣΑ να ακολουθήσουν και να συμμορφωθούν με τις συστάσεις του και εγχωρίως και εξωτερικά για το πώς ε, αναθεωρούν, προσαρμόζουν και ερμηνεύουν τις συμφωνίες τους με άλλες Αλλά το θέμα είναι πώς θα επιβληθεί και ε, ο σχετικός νόμος από τις σχετικές αρχές. Είναι κάτι που θα χρειαστεί πολύ χρόνο και πολλοί από τις υπευθύνους θα έχουν εκτίσει και την ποινή φυλάκισή τους μέχρι να ολοκληρωθεί το σύστημα. Η ερώτηση των εισηγητών είναι τι μπορεί να κάνει εδώ το Ευρωκοινοβούλιο. Τι μπορεί να γίνει εντός της Ευρώπης. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, να πω ότι είναι τουλάχιστον τρεις τομείς που μπορείτε να δράσετε. Πρώτον, όπως είπε ο Έντουαρτ, ο Εντουάρ, θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προστασία για τους καταγγέλλοντες. Αυτούς που προστατεύονται που προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον και δεν καταγγέλουν μόνο και μόνο κάτι παράνομο. Ε, κάποιοι είναι εξαιρετικά θερά, λέει, ότι πρέπει να υπάρχει επίση μεγαλύτερη διαφάνεια για τι φορολογικέ συμφωνίε εντό Ευρώπη. Θα πρέπει να είναι τελείω ε, δημόσιε. Με, κατονομα... με τι εταιρείε να κατονομάζονται εφόσον αυτό γίνεται. Και εφόσον δεν υπάρχει ακόμα μια πλήρη λύση από τον ΩΣΑ για το θέμα της φοροαποφυγής, θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσει από το ευρωπαϊκό επίπεδο για όσου εκμεταλλεύονται την ελευθερία που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκέ συνθήκε, για να εξαπατήσουν στην ουσία άλλα κράτη-μέλη και άλλε ευρωπαϊκέ εταιρείε. Οι κυρώσει αυτέ θα μπορούσαν να είναι ακριβώ φορολογικέ. Δηλαδή να μπορεί κανεί ελεύθερα να βάζει και να βγάζει το χρήμα, τα χρήματά του στο Λουξεμβούργο όπω θέλει. Χωρίς επιβολή κανένας φόρου. Υπάρχουν λοιπόν μερικά άμεσα μέτρα που μπορεί να, να ληφθούν. Αλλά δεν υπάρχει τέλεια πολιτική λύση. Μόνο η απόλυτη διαφάνεια είναι η άριστη κατεύθυνση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ συγκεκριμένε συστάσεις. Νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν λέτε ότι υπάρχουν δύο επίπεδα δράσης που ανοίγονται. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δράσουμε και στα δύο επίπεδα. Το παγκόσμιο, βάσει των συστάσεων του ΩΣΑ, και το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν εδώ ιδιαίτερα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να είναι ένας χώρος αλληλεγγύης. Εάν αφήσουμε χωρίς έλεγχο ένα σύστημα όπου κάποιοι κλέβουν φορολογικά έσοδα από άλλους, για όλου του λόγου οπότε αυτό δεν είναι θεμητό, αλλά εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη σκοπιά τη αλληλεγγύη έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι και κάπω ε, διαφορετικό σε σχέση με το τι συμβαίνει στην κλίμακα την διεθνή. Τώρα, οι εκπρόσωποι των ομάδων έχετε δύο λεπτά καθένα για τι ερωτήσει και τα σχόλιά σα και μετά θα μπορέσετε να απαντήσετε. όπως θα το θελήσετε, ε, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Έγγελ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω λέγοντας ότι οπουδήποτε οι δημοσιογράφοι διώκονται επειδή κάνουν τη δουλειά τους, αυτό δεν δείχνει καμιά ιδιαίτερη πολιτική ή δικαστική ευφυΐα. Λυπούμε πάρα πολύ. Βρώ τη λύπη μου που κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Αν και δεν εκφράζω τη λύπη μου ιδιαίτερα αναφορικά με ό,τι είπαν ορισμένοι, ότι κανείς παραβιάζει τον νόμο αποκαλύπτοντας πληροφορίες που δεν απευθύνονται στο κοινό. Δεν μπορεί ωστόσο το δικαστικό σύστημα να κάνει σαν να μην συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Βρίσκω ανόητο λοιπόν να διώκονται δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν στην πραγματικότητα τη δουλειά τους. Θεωρώντας, έστω και υποκειμενικά, ότι υπερασπίζεται το δημόσιο δίκαιο, τα δικαιώματα του κοινού. Όλα αυτά τέλος πάντων δεν μπορεί ωστόσο να σταματήσει κανείς σε αυτά, ούτε εσείς ούτε εμείς εγώ θα ήθελα να γνωρίζω εάν μέσα στο πλαίσιο που έχουμε σε παγκόσμια κλίμακα, δηλαδή έναν άγριο ανταγωνισμό για την προσέλκυση των εδρών των διεθνών, μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων. Αν λοιπόν υπάρχουν ενδεχόμενα κάποιες προτάσεις πιο ελκυστικές από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα ώστε στην Ευρώπη κλείνοντας κάποια χρηματοπιστωτικά κέντρα να χάσουμε και τις επιχειρήσεις. Ούτε πιστεύει κανένα ότι όλοι θα πάνε σαν γκάι βέβαια. Αλλά θέλω να μάθω ποια βήματα, ποια κοινά διαβήματα μπορούμε να κάνουμε, να αναλάβουμε ώστε ενδεχομένως και προς όφελος ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στον τομέα αυτό και ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις μια ηθική στάση και μια ηθική υποχρέωση να παραμείνουν στην Ευρώπη και να διατηρήσουν την Ευρώπη ως έδρα τους έστω και αν κληθούν τελικά να πληρώνουν κάτι παραπάνω από ό,τι πληρώνουν σήμερα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Τώρα εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Σκόφοντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριοι για τις ε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σας. Πρώτα θα ήθελα να πω στον κύριο Περίν ότι το γεγονό και μόνο ότι το Λουξεμβούργο σας διώκει για τις διαρροές για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε να είναι αδύνατον. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα κανόνα που να λέει ότι αν για παράδειγμα η Κομισιόν και αυτοί τώρα διεξάγουν έρευνα εφόσον το πράτη κάνει μια διαρεύνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει όσο υπάρχει τέτοια έρευνα να μπορεί μια χώρα να στρέφεται κατά των δημοσιογράφων. Είναι απόλυτα παράδειγμα λοιπόν που το Λουξεμβούργο προβαίνει σε δίωξη σε βάρος Αυτό είναι πραγματική επίθεση κατά της ελευθερίας του τύπου και παραβιάζει τις αξίες μας, του κράτους δικαίου, τη αποκάλυψή παραβιάσεων στι οποίες προβαίνουν οι αρχέ. Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες ώστε στο μέλλον να είναι απολύτω αδύνατο κάτι τέτοιο. Όταν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά μια συγκεκριμένη υπόθεση να μην μπορεί η χώρα μέλο να προβαίνει σε δίωξη κατά των δημοσιογράφων που έχουν αποκαλύψει την υπόθεση. Δεύτερο, θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους καταγγέλλοντες και τα άτομα δηλαδή που χρησιμοποιείτε εσεί ενδεχομένω ως πηγές ή που εργάζονται και μέσα σε θεσμούς. Έχετε τίποτε καλέ ιδέε για το πώ να του προστατεύσουμε. Επίση, τι κίνητρα μπορούμε να προσφέρουμε σε καταγγέλλοντες για να προβούν στις αποκαλύψεις των πληροφοριών που κατέχουν. Από την δική σας εμπειρία τι προκύπτει. Δεύτερο, απευθυνόμενος ίδιος τον κύριο Μπρούξ. Είπατε κάτι ουσιώδες στη συζήτηση αυτή. Μια από τις χώρες που περιγράψατε, το Λουξεμβούργο, είναι πλήρε μέλος των θεσμικών οργάνων όπου βρισκόμαστε και εμείς και βεβαίω χαίρουν τη προστασία που χαίρουν οι χώρε μέλη και τη προστασία από την συνθήκη. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω να επεκταθείτε λίγο περισσότερο. Τι είδους κυρώσει θεωρείτε ή τέλος πάντων τι είδους οδοί οδηγούν σε κυρώσεις και χρησιμοποιεί το Λουξεμβούργο την θέση του για να μπορεί να επιβάλλει τις πρακτικές αυτές που βοηθούν τις εταιρείε να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και στην ουσία είναι δηλαδή εγκληματικέ πράξεις. Όταν δηλαδή τη διευκολύνει το Λουξεμβούργο να μην πληρώνει φόρους εκεί όπου προκύπτει το κέρδος των επιχειρήσεων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Για την τελευταία σας ερώτηση μάλλον εμείς είμαστε πρέπει να απαντήσουμε. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές ο κύριος Κλαστοντέσκη, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω πολωνικά, αν με επιτρέπετε. Because I could also in Θα μπορούσα και γερμανικά ή αγγλικά, αλλά είναι και αυτή η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρόεδρε, θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, δημοσιογράφους μας για την ερευνητική τους δουλειά και να τονίσω το ρόλο τους για τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, τις δημοκρατικές αρχές. Είναι θεμελιώδης η λειτουργία που εκτελούν. Όμως, ακούγοντας και όσα είπαν συνάδελφοι, να πω το εξής. Ίσως να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή κρίση στην ερευνητική δημοσιογραφία, διότι δόθηκε το παράδειγμα ποινικών ε, διώξεων. Δεν είναι περίεργο αυτό διότι υπάρχουν πολλές καταστάσεις όπου αντιμετωπίζουμε το ίδιο φαινόμενο. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξής. Εάν μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την πίεση που έχετε υποστεί. Ε, είναι σημαντικό αυτό για τις ελευθερίες ε, των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης και τα κλασικά μέσα πάνω απ' όλα. Και επίσης ερώτημα για την ερευνητική δημοσιογραφία γενικότερα. Θα πρέπει την ερώτηση αυτή να την δούμε πολύ σοβαρά και στο Κοινοβούλιο. Την έκανε και ο Μιχαήλ Τόιρεφ την ερώτηση για τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δεν είναι απλώς υπεύθυνα για τα δικήματα ή τα εγκλήματα αυτά, αλλά και πολλές φορές και θύματα, διότι οι πιο αδύναμοι δεν μπορούν να προστατευτούν έναντι της ε, παντοδυναμίας των πολυεθνικών. Ίσως λοιπόν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να ε, επιτείνει την ε, ευάλωτη αυτή θέση κάποιων κατών μελών σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Όχι μόνο να καταδικάζουμε αυτές τις πρακτικές, ακόμη και αν είναι νομότυπες ε, ή νόμιμες τυπικά αλλά νύφικες. Σε κάθε περίπτωση προσεκτείουν τα κεφάλαια των επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να δούμε και την ευάλωτη θέση κάποιων χωρών εναντί του κεφαλαίου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Φανίβενχόιζεν. Από του φιλελευθέρου, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά κι εγώ τη σειρά μου. Ε, σας αφήνω λίγη ε, ώρα να βάλετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ πολύ τους δημοσιογράφους που ήρθατε εδώ. Ε, ήταν πολύ εντυπωσιακά αυτά που μας είπαν ε, και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τον όγκο που έχουν αποκαλύψει. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία να αναμένουμε. Γιατί ε, στο LuxLeaks συνήθως συζητάμε για τα rulings. Αλλά εμείς έχουμε ως εντολή στην Επιτροπή μας να το ψάξουμε περισσότερο ε, για να δούμε και άλλα θέματα που μοιάζουν με αυτές τις φορολογικές συμφωνίες. Έχετε στη δική σας έρευνα ε, βρει τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχουν άλλου είδους κρατικές ενισχύσεις για να το πω έτσι, συμφωνίες όχι μόνο για φορολογικά κίνητρα αλλά και για επιδοτήσεις, κρατικές ενισχύσεις σε τέτοιου είδους εταιρείε με πλάγιους τρόπους και θα ήθελα να το συνδέσω και με κάτι άλλο. Πολύ συχνά ε, επικεντρωνόμαστε σε αμερικανικές εταιρείες, ε, αλλά ο κόσμος είναι περίπλοκος και είναι και διεθνής. Ε, τι λένε οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, και από την Αμερική συνεργάζεται με αυτούς. Πώς το βλέπουν με Αυστραλούς, από ό,τι κατάλαβα, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα θέματα τα φορολογικά, ακόμα και η Κίνα ασχολείται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς έχουν οι επαφές σας με τους συναδέλφους σας διεθνώς και να το συνδέσω και με κάτι άλλο. Συνέχεια μιλάμε για εταιρείε, για επιχειρήσει, αλλά όλο και περισσότερο ακούμε και για μη κυβερνητικέ οργανώσει που παίρνουν λεφτά για αναπτυξιακή βοήθεια και τα διοχετεύουν σε συγκεκριμένες χώρες με διάφορα ε, κατασκευάσματα και φορολογικούς παραδείσους. Και δεν φτάνουν τα λεφτά στους τελικούς δικαιούχους, δεν τους τα δίνουν, λέει, γιατί είναι ε, διεφθαρμένα τα καθεστώτα. Αυτά τα έχετε αντιμετωπίσει, τα έχετε δει και τι κάνετε σχετικά. Έχω και άλλη ερώτηση, χρόνο δεν έχω κρίμα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κόρα. Από την Ενωτική Αριστερά, ο Φάβιο Δημάζη. Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ όλους προσκεκλημένους ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ και τον Μίχαελ Τόιρερ για τη διευκρίνηση προηγουμένως. Έχω την εντύπωση ότι εδώ μέσα καμιά φορά η ε, πλειοψηφία δεν ενδιαφέρεται περισσότερο να προστατεύσει τους δημοσιογράφους ή τους καταγγέλλοντες, αλλά τον κύριο Γιούνκερ. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω επίση ότι λυπάμαι και εγώ κύριε Περέ που δεν είμαστε εμεί διερευνητική εξεταστική επιτροπή και επίση λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να φέρουμε εδώ τον κύριο Ντελτούρ. Θα ήθελα να προσθέσω όμω το εξή μόνο. Οι αποκαλύψει του κυρίου Περάν και κάποιων άλλων ε, αποκαλύψει νομίμων δραστηριοτήτων θα πρέπει να το μελετήσουμε γιατί υπάρχει μια εγκύκλειος του 1989 ε, της εφορίας του Λουξεμβούργου ε, που λέει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ε, τις δυνατότητες που έχουν για φορολογική βελτιστοποίηση ορισμένοι. Ακόμα και αν υπάρχει ένα τέλμα φορολογικό. Είναι περίεργο λοιπόν που ασκούν ποινική δίωξη στον κύριο Πέρα που αποκαλύπτει κάποια πράγματα. Ελπίζω να βρεθεί εδώ πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για την οδηγία για την προστασία του εμπορικού απορρίτου. Να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Περάν κυρίως, αν θεωρεί ότι αυτά που έχει εξαγγείλει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών για τα φορολογικά σημειώματα ή τις φορολογικές δηλώσεις και ε, συμφωνίες μάλλον, ε, το θεωρείτε λογικό ε, σκόπιμο και οι συστάσεις, οι εκθέσεις αναχώρα θα πρέπει να είναι δημόσιες και τελικά περιμένετε και για καταγγέλλοντες και για δημοσιογράφους να υπάρχει δυνατότητα μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Safe Clouds και τα λοιπά να διαβιβάζουν τις πληροφορίες τους για να μην καταλήγουν πάντα στο εδόλιο του κατηγορουμένου αλλά μπορέσουμε και εμείς κάπως να τους προστατεύσουμε. Ευχαριστώ από τους Πρασίνους η κυρία Εύα Ζολή, Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσει. Η πρώτη, στον κύριο Περά. Κύριε Περά, στις έρευνέ σα, τι ε, συζητήσεις είχατε με τους αρχέ του Λουξεμβούργου, τι στάση τήρησαν και τι επίπεδο διαφάνειας και συνεργασία ε, φάνηκε να έχουν. Ε, έπειτα προς όλους τους προσκεκλημένου, ο κύριος Πέρα πρόσφατα ε, προσήχθη ενώπιον της ε, δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου, κυρίως για την παραβίαση του εμπορικού απορρίτου. Πιστεύετε ότι μια τέτοια ε, δίωξη θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλο κράτος Πιστεύετε ότι το έργο αυτής της ειδική Επιτροπής συνάδει με το σχέδιο οδηγίας για το απόρριτο των εμπορικών υποθέσεων και εάν ισχύουν όσα μαθαίνουμε ε, από τα μέσα, η οδηγία αυτή προωθήθηκε από πέντε πολυεθνικές και τρεις ε, ομάδες πίεσης ε, εσάς ε, σας ε, απευθύνθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η η συγγητρια της για το θέμα αυτό. Merci, Ευχαριστούμε κυρία Ζολή για την Ευρώπη της Δημοκρατία και ο κύριος Βάλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους που ήρθαν εδώ για το διάλογό μας και τους ευχαριστώ για το θάρρος τους, την πνευματική τους διάβγεια και την ε, λογική που δείχνουν σε όλο, αυτή, αυτόν τον αγώνα κατά του τεράστιου συστήματος αυτού και του παράλογου που πρέπει να καταπολεμήσουμε με τις πολυεθνικές που ακόμη και σήμερα μπορούν να μετακινήσουν ε, ποσά όπως θέλουν με τεράστιους φορολογικούς ελιγμούς στις χώρες του G8. πρέπει να ξαναδούμε τη χάραξη ολόκληρης της φορολογικής πολιτικής. Ήθελα τη γνώμη σας για την πολύ στήρα στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πόσο πιστεύετε ότι η Επιτροπή Juncker θα πετύχει να κάνει κάτι παραπάνω χειροπιαστό, ε, τι χειροπιαστά μέτρα θα μπορούσε να λάβει για να εξαλείψει το πρόβλημα αυτό. Ε, η πιθανότητα των κυρώσεων ε, ήδη ακούστηκαν από την πλευρά του ΟΣΑ. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε αυτό το σύστημα να λειτουργήσει ε, από τον πολιτικό χώρο για να επιβληθούν επιτέλους και κάποιες κυρώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους μη εγγεγραμμένους. Ο κύριος Ζαριανόπουλος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, για την πρώτη ερώτηση που ήθελα να θέσω δημοσιογράφους έχω πάρει ήδη απάντηση ήταν για το θέμα των διώξεων εναντίον τους και των επιπτώσεων. Ωστόσο να σημειώσω ότι οι διώξεις κατά των καταγγελόντων και όσων αποκαλύπτουν ε, δείχνουν και το περιεχόμενο και την ουσία της δημοκρατίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη ποιος τελικά ασκεί την πραγματική εξουσία. Ένα ε, δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να απευθύνω είναι το εξή. Αν ε, μετά την έρευνα που κάνουν θεωρούν ότι υπάρχει περίπτωση να δοθεί έστω κάποια λύση αν δεν αρθεί ολοκληρωτικά το τραπεζικό και το φορολογικό απόρριτο σε όλες ε, στα κράτη-μέλη. Και τελευταίο. Την προηγούμενη φορά είχαμε προσκαλεσμένες τις τέσσερις μεγάλες διεθνείς ε, εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμβουλών. Είχα απευθύνει εκεί μια ερώτηση, είχα δηλώσει ότι δεν περίμενα απάντηση, γιατί αν δίναν απάντηση θα ήταν σαν να ε, αναιρούν την ίδια τους την ύπαρξη, ω εργαλεία αυτής της πολιτικής της φοροαποφυγής. Ωστόσο, θα ήθελα στου ερευνητέ δημοσιογράφου να απευθύνω την ίδια ερώτηση, μια και έχουν κάνει έρευνα και μάλιστα χρήσιμη, έχουν κάνει διαπιστώσει και έχουν δει τι προποθέσει και τι υποδομέ που, που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, η ερώτηση είναι η εξή. Βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελευθερία κίνησης κεφαλαίου. Μέσα σε αυτή την ελευθερία, αξιοποιώντας την, αυτή την τεχνική, ας το πούμε, οικονομική δυνατότητα, κεφάλαια διακινήθηκαν προς φορολογικούς παραδείσους. Δεύτερον, βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρεί ως κινητήρια δύναμη αυτά τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα είναι ότι πρέπει να τους δοθούν κίνητρα μεταξύ των οποίων και, φοροαπο... και μείωση φορολογικών συντελεστών, δηλαδή φοροαποφυγή ουσιαστικά νόμιμη. Αυτό είναι το πολιτικό περιβάλλον. Αυτό περιγράφεται και σε όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θεωρούν ότι μπορούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της φοροαπαφυγής που τελικά είναι νόμιμη. Ε, σε διάφορες χώρες και συνολικά στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δηλαδή πρόβλημα νοοτροπίας κάποιων κακών πολιεθνικών, είναι πρόβλημα τεχνικών αδυναμιών της Ένωσης και των κρατών μελών της ή τελικά, όπως πιστεύουμε εμείς, είναι ζήτημα της φύσης του ίδιου αυτού του οικονομικού συστήματος το οποίο υπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτήν. σε πολύ. Θα προσεθετά εγώ ίδιος με παρατηρήσει και μερικές ερωτήσεις. Πρώτα, να, ενημερώσουμε την ομιγυρία για τους προσκεκλημένους μας ότι Ήδη σε έξι χώρες κατά τη μέλη περίπου έχουμε οργανώσει επισκέψεις για ενημέρωση. Σήμερα ε, θα κάνουμε τη σχετική επίσκεψη εδώ στο Βέλγιο με τις βελγικές αρχές και την επόμενη εβδομάδα έχουμε προγραμματίσει το Λουξεμβούργο. Ε, οι συνάδελφοι από το Λουξεμβούργο ξέρουν, όπω ο κύριο Έγγελ, ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μα για να συλλέξουμε πληροφορίε και εκεί. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις μου. Οι πρώτες έρευνες που έσπασαν το φράγμα της αδιαφορίας, ένα πραγματικό τείχος αδιαφορίας της κοινή γνώμης, ξεκίνησαν ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ένας δημοσιογράφος της New York Times πήρε το βραβείο Pulitzer για μια τέτοια έρευνα. Εγώ πήγα στη χώρα αυτή και συνάντησα γερουσιαστές που είχαν διοργανώσει πολύ ενδιαφέρουσες ακροάσεις όπως η σημερινή ε, η δική μας και αυτές που έχουμε οργανώσει ε, αναλόγως εδώ και κάποιες εβδομάδε, και την εποχή εκείνη υπήρχε μια πραγματική πολιτική διάθεση και βούληση να δώσουν τέρμα σε μια κατάσταση που όλοι τη θεωρούσαν ε, κάτι που ήταν πραγματικά συγκλονιστικό και τρομακτικό. Ε, αυτή η πολιτική βούληση δεν υπάρχει πια. Ε, πώς θα ξαναβρούμε αυτή την πολιτική όθηση εάν δεν υπάρχει συνολική, ε, ομαδική ε, διάθεση από τα μέλη μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πληροφοριών που αυτά μπορούν να παράσχουν με την ισορροπία, με την έχοντα υπόψη μόνο ότι οι αρμοδιότητε του Ευρωκοινοβουλίου δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν την έλλειψη δράση από πλευρά των 100 μελών. Από αυτήν την σκοπιά. Θα θέσω ένα ερώτημα στο οποίο μπορείτε να μην, να μην απαντήσετε βεβαίω, γιατί σα δεσμεύει το επαγγελματικό σα απόρριτο. Αλλά δεν θα σα κατηγορήσει κανεί γι' αυτό. Μετά την έρευνα για το Λουξεμβούργο. Έγιναν έρευνε και για την Ελβετία. Και είναι σαφές ότι δεν είναι μόνο οι χώρες αυτές στην Ένωση ή στο περιθωριό της που δημιουργούν προβλήματα και των οποίων το νομικό σύστημα, οι φορολογικές αρχές επιτρέπουν αυτό που θα ονομάζαμε από νομικής πλευράς φόρο αποφυγή. Έχετε σκοπό να προχωρήσετε και σε επιπλέον έρευνες. Η δική μου η αίσθηση υπερβάλλοντας ίσως κάπως, είναι, για να κάνω και μια παρομοίωση, είναι ότι στους κόλπους της Ένωσης κάθε μια από τις 28 χώρες είναι ο φορολογικός παράδεισος κάποιες άλλες. Υπάρχουν κάποιοι πιο πολυτελείς παράδεισοι, πιο ε, γενναιόδοροι οικοδεσπότες από άλλους, αλλά την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία όταν ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σαπά, ήρθε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, να του θυμίσω ότι, ότι χάρη στην ε, France 2, αυτό το κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης, έχουμε δει ότι εταιρείε που ελέγχονται από το γαλλικό κράτος, όπως η Aeroport de Paris, η EDF, η Renault, έχουν αξιοποιήσει μέσα φορολογικής βελτιστοποίησης που θα ήταν αρκετά περίεργα και θα ευνηδίαζαν αν τα γνώριζαν οι πολίτες. Ήταν μάλιστα μια ευκαιρία το Υπουργείο Οικονομικό να λάβει μέτρα και να δώσει τέλος σε αυτές τις περιπτώσεις και μάλιστα σε, όχι μόνο για εταιρείες στην γαλλική επικράτεια, αλλά και σε κράτη όπου οι γαλλικές αυτές εταιρείες είχαν παρουσία. Αυτά για το πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύσει διαφορετικά το, ε, το γράμμα του νόμου. Και ήθελα να σας προειδοποιήσω ε, σας τους δημοσιογράφους ή μάλλον να ζητήσω από σας την συμβουλή σας δάση της πείρας σας. στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα έχουμε ακούσει αρκετέ φορέ στην Ολομέλεια και μάλιστα νομίζω ότι σε επίπεδο πλειοψηφία έχει υποθεί αυτό. Εάν υπήρξε, αν υπάρχει δυνατότητα για ένα σύστημα προστασία μαρτύρων σε αυτή την περίπτωση. Νομίζετε ότι είναι κάτι που το δικαιούνται οι πηγέ των δημοσιογράφων, προστασία των πηγών δηλαδή των δημοσιογράφων. Ή μήπω υπάρχει μια διάσταση που ξεπερνά απλώς τη λειτουργία αυτή το να είναι κανείς πηγή για δημοσιογράφους. Είναι το ίδιο πρόβλημα ή κάτι διαφορετικό, κάτι παράλληλο. Σας ευχαριστώ και απαντήστε με όποια σειρά θέλετε. Κύριε Σπέρα, ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις θα απαντάμε ένας μετά τον άλλον. Θα ήθελα να επανέλθω σε διάφορα θέματα που αναφέρατε εσείς ο ίδιος Πρόεδρε, αρχίσω από το τέλος. Γιατί το φράγμα της αδιαφορίας που έσπασε πριν από λίγα χρόνια ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε μετά από μια προσπάθεια που έχει χαθεί αυτή η όθηση. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να ε, ξυπνήσει ο κόσμος να αρχίσει να ενδιαφέρεται με έρευνες. Θυμίζουμε ότι ακόμα υπάρχουν τα ίδια διακυβεύματα και απέναντί μας είναι κάποιοι πάρα πολύ ισχυροί που έχουν τον τρόπο τους για να προωθούν τη δική τους ατζέντα και τα δικά τους θέματα και, να καθορίζουν και το χρονοδιάγραμμα και την πορεία, την ταχύτητα των πραγμάτων. Ε, επανειλημμένα ε, μας ρωτήσατε πού θα ερευνήσετε, σε ποιο αντικείμενο. Ε, θα απαντήσω προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και οι συνάδελφοι το ίδιο, ε, ότι δεν θα επεκταθούμε αυτή τη στιγμή σε αυτό, θα δείξει. Επίσης, ε, μας ρωτήσατε τι έχουμε να σας πούμε για την επικείμενη επίσκεψή σας στο Λουξεμβούργο. Θα ζητήσετε να ακούσετε τον κύριο Μάριους Κόλ. Βλέπετε αυτό στο Λουξεμβούργο. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα σας πει για την ταχύτητα με την οποία εργάζεται και τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, ε, τσέκαρε τις πληροφορίες που είχαμε για τα, τις φορολογικές συμφωνίες αυτές. Θέλω να επανέλθω λίγο στο θέμα της προστασίας των πηγών και των καταγγελόντων. Η πρώτη φάση για μένα, το πρώτο στάδιο θα ήταν να υπάρχει μια συνοχή στη δουλειά τι συμβαίνει εδώ και τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδηγία σχετικά με το εμπορικό απόρριτο. Το είπα από την αρχή αυτό. Δεν υπήρξε προηγούμενη διαβούλευση για το σχέδιο οδηγίας. Εγώ το θέμα το γνωρίζω προσωπικά αρκετά καλά, διότι ε, στο δικό μου ε, πρακτορείο ήμασταν αρκετοί από το ε, Ιανουάριο και στραφήκαμε κατά ενός αντίστοιχου νομοσχεδίου για την παραβίαση του εμπορικού απορρίτου στη Γαλλία. Καταφέραμε να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο γιατί ξέραμε ότι στη συνέχεια ακολουθούσε μια ευρωπαϊκή οδηγία. Ε, με ρωτήσατε αν είχαμε επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Σας απαντώ όχι. Εμείς το ανακοινήσαμε. Εμείς ε, απευθυνθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ήρθε κανένα σε επαφή μαζί μας, ούτε μας ρώτησαν προηγουμένως, ούτε επεδίωξαν να μα συναντήσουν. Απαντώ στην κυρία Ζολή για την συμπεριφορά της κυβέρνηση του Λουξεμβούργου και των αρχών γέννη σε ό,τι με αφορά κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου ήταν πάντα φαινομενικά ευγενής μας είπαν ότι έχουμε φόρο εταιρικό 29 και κάτι της 100, σεβόμαστε τον νόμο και δεν έχουμε ε, τίποτα επιλήψιμο κάνει. Και το λέω και στους συναδέλφους, δεν ξέρω αν είχαν την ίδια αντιμετώπιση, εμένα αυτή την αντιμετώπιση μου επιφύλαξαν ε, συνεχώς. Τώρα, για το θέμα του εμπορικού απορρίτου είναι ένα μείζον ζήτημα και πρώτα απ' όλα είναι πρωταρχικό να υπάρχει μια συνοχή ε, στα όσα κάνετε εσείς και αυτά που προτίθεται να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Και μόνο το γεγονό ότι μπορεί κανεί να απειλήσει προδικαστικά χωρί να κινηθεί καμία διαδικασία μπορεί να σταματήσει τι έρευνε ε, σε εμβρικό στάδιο. Δηλαδή αρκεί κάποιε εταιρείε να στείλουν ε, ε, κάποιες επιστολές από δικηγορικά γραφεία για να κάνει πίσω ο δημοσιογράφος και να μην συνεχίσει την έρευνα. Θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου, ο κύριος Μποβέ τώρα. Μποβέ. Είστε συγγενείς του συναδέλφου μας, Ζε Μποβέ. Ε, όχι, όχι. Όχι. Ξέρω, σας καθησυχάζω. Ε, προσωπική ήταν η ερώτηση αυτή. Όχι, όχι, σας ε, καθησυχάζω. Καμία σχέση. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω Ολλανδικά βεβαίως μπορείτε. Νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση ε, ήταν η κεντρική ιδέα του προβλήματος, αν είναι νόμιμο αυτό ή όχι. Και πραγματικά εδώ βρισκόμαστε στην ουσία του προβλήματος. Γιατί, διότι μπορώ να σας δώσω παραδείγματα από το Βέλγιο, γιατί εγώ είμαι Βέλγος, θα πρέπει ήδη να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στο ότι είναι ποινικά νόμιμο και τι είναι διοικητικά νόμιμο ή φορολογικά εντάξει. Αυτές είναι οι δύο διαφορές. Και μπορώ να σας πω ήδη από την αρχή ότι έγιναν έρευνες και διαπιστώθηκε ότι ορισμένα κατασκευάσματα ε, είναι, αγγίζουν την ε, ε, απάτη την πλαστογράφηση δηλαδή, αλλά ε, ε, τα άλλα θέματα, τα διοικητικά, είναι πολύ περισσότερα ε, απέναντι στα ποινικά και είναι φορολογικά κατασκευάσματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα να τα δεις αυτά. Στο Βέλγιο, πριν από το LuxLeaks, είχαμε πολλές περιπτώσεις όπου προσπάθησε η εφορία, η επιθεώρηση της εφορίας, να ε, στιγματίσει εταιρείες θηρίδες που πραγματικά έχουν δημιουργηθεί μόνο ε, στο Λουξεμβούργο για να ε, φοροδιαφεύγουν. Προσπάθησε λοιπόν η εφορία να τους πιάσει και να ζητήσει τα φορολογικά έσοδα που διέφευγαν και αυτή ήταν και μια ε, μεγαλύτερη ε, εταιρεία τηλεπικοινωνιών που είναι σε μεγάλο μέρος ιδιοκτησία του κράτους και μια πολύ μεγάλη ε, γαλλική ενεργειακή εταιρεία. Και τις δύο περιπτώσεις τις έχασε η βελγική εφορία και έρχομαι σε αυτό το θέμα της ουσίας. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε όσους κανόνες θέλουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, αλλά πότε έχει ε, κάτι ε, πώς να το πω, ουσιαστική ε, υπόσταση. Πότε μια εταιρεία που εδρεύει στο Λουξεμβούργο χαρακτηρίζεται θηρίδα μαϊμού και πότε είναι holding. Αυτό δεν μπορείς εύκολα να το αποδείξεις. Ε, υπάρχει ας πούμε μια διεύθυνση στο Λουξεμβούργο που εδρεύουν εκατοντάδες εταιρείες και νοικιάζουν απλώς τη διεύθυνση. Ε, δηλαδή αν είχαν νοικιάσει ένα μεγαλύτερο γραφείο και όχι μόνο την ταχυδρομική θηρίδα θα ήταν νόμιμα. Δηλαδή πού βρίσκεται η ουσία είναι δύσκολο να το αποδείξεις η οικονομική. Όλα αυτά τα κατασκευάσματα που μελετήσαμε με τα ε, Lux Leaks είναι ότι είναι δύσκολο αυτό να αποδειχθεί. Δεν υπάρχει οικονομική ουσία, ε, δεν υπάρχει πραγματική οικονομία παρά μόνο φορολογική σκοπιμότητα. Αυτός ήταν ο λόγος ύπαρξης και κανένα άλλος. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να ψάχνουμε την οικονομική ουσία πίσω από αυτά τα κατασκευάσματα για να βλέπουμε τι ευσταθεί και τι όχι. Ένα άλλο στοιχείο είναι η διαφάνεια. Τα rulings, αυτές οι συμφωνίες μπορεί να είναι καλό σύστημα, αλλά οι λουξεμβουριανές αρχές έχουν κάνει απόλυτη κατάχρηση σε τεράστια κλίμακα. Δίνουν σε εταιρείε δυνατότητες να ερμηνεύουν διάφορα πράγματα και διάφορους φορολογικούς νόμους για να έχουν πλήρη ασφάλεια ε, κατέστη δυνατό να πάρουν το πράσινο φως για να ε, κατασκευάσουν ε, διάφορα εφάνταστα ε, και να είναι και μια πύλη εισόδου προς πραγματικούς φορολογικούς παραδείσους. Έτσι η πιο πλούσια βελγική οικογένεια έστειλε στο Γιβραλτάρ μερίσματα εκατομμυρίων ευρώ και αν δεν υπήρχε το LuxLeaks η εφορία δεν θα έπαιρνε μυρωδιά. Διότι είπαν ότι ήταν μια holding από το ε, Λουξεμβούργο και πήρε το OK, το Fiat με την ε, συμφωνία, ε, το ruling του Λουξεμβούργου. Επίσης υπάρχουν και κάποιες επιτροπές για αυτές τις συμφωνίες, rulings, που έχουν μια τεράστια ελευθερία για να δίνουν το πράσινο φως για διάφορα τέτοια είδους κατασκευάσματα. Και εμείς διαπιστώσαμε ότι ακόμα και η νομοθεσία που υπάρχει στο Λουξεμβούργο, ας πούμε, για την πνευματική ιδιοκτησία, όπου ε, ε, υπάρχει 80% φοροαπαλλαγή. Ε, υπάρχει και στο Βέλγιο αυτό, αλλά η δική μας Επιτροπή για τα rulings έχει πολύ πιο αυστηρή και περιοριστική ερμηνεία από τη διευρυμένη που έχουν στο Λουξεμβούργο. Δηλαδή, ε, όταν έχεις μια βελγική ε, εταιρεία με πνευματική ιδιοκτησία, ε, απερίφθη από τη Βελγική Επιτροπή και πήγε στο Λουξεμβούργο που τους το ενέκρινε. Και το κατασκεύασμα που τους εγκρίνανε κάπως ερμήνευε ελαστικά την ίδια την νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει έλεγχος και στις επιτροπές που κάνουν αυτές τις συμφωνίες. Αυτό γίνεται και με διαφάνεια αλλά και με τις εθνικές κυβερνήσεις που είναι υπεράνω. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι κάθε χώρα φέρει την ευθύνη για τους φορολογικούς του νόμους προφανώς και κάθε χώρα έχει παραθυράκια σαφέστατα στις νομοθεσίες αυτές όπου στο Λουξεμβούργο όταν τα ε, ε, διαπίστωσαν ότι υπάρχουν έχουν κάνει τρομερή κατάχρηση. Ε, στο Βέλγιο υπάρχει ένα σύστημα BEVEX που είναι ένα σύστημα επενδυτικό για να μην επεκταθώ. Στην πρώτη φάση δεν φορολογείται, στη δεύτερη φάση φορολογείται. Έχτισαν λοιπόν ένα σύστημα, άμα πας στο Λουξεμβούργο και είσαι στην πρώτη φάση Κάνεις την πρώτη φάση στο Βέλγιο, μετά πας στη δεύτερη φάση στο Λουξεμβούργο, έχεις ευνοϊκό καθεστώς για τα holding, άρα μηδέν φορολογία. Ε, δηλαδή έτσι αξιοποιούν τη βελγική νομοθεσία και μετά πηγαίνουν στο Λουξεμβούργο. Και αυτό δεν γίνεται σε περιορισμένη μικρή κλίμακα, αλλά ε, έγινε λόγος για πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις ε, που γίνονται ε, με μηδενική φορολογία. Και επίσης οι ίδιοι οι δικαστές στο Λουξεμβούργο επιτέλους και τελικά έδεισαν την έγκρισή τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο η νομοθεσία, είναι και πώς εφαρμόζεται και η δικαιοσύνη πρέπει να κλείσουν αυτά τα παραθυράκια. Ναι. Ε, Ευχαριστώ κύριε Κλέριξ. Και εγώ θα μιλήσω Ολλανδικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ σε αυτή την ακρόαση για να σας δώσουμε περισσότερες διευκρινήσεις. Ε, χαίρομαι που πήρε τέτοια διάσταση το θέμα των LuxLeaks και δόθηκε αυτή η συνέχεια. Μπορώ να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Η κυρία Φερέιρα ρώτησε αν έχουμε ε, δημοσιεύσει τα περισσότερα στοιχεία ή αν έχουμε και άλλα προς δημοσίευση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μετά ε, την πρώτη δημοσίευση Offshore Leaks, Lux Leaks και Swiss Leaks. Ε, ο Διεθνής Όμιλος ε, Ερευνητών Δημοσιογράφων κινητοποιεί όλο και περισσότερους καταγγέλλοντες που έρχονται και κρούν το κόδωνα του κινδύνου αλλά και τις δικές μας θύρες με πληροφορίες. Με τον τρόπο που λειτουργεί στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, μέσω δημοσιογραφικής έρευνας. Και αυτό είναι και το πλεονέκτημα. Έχουμε μια παγκόσμια οργάνωση και είμαστε μοναδικός παραλήπτης. Ε, οπότε ε, βεβαίως η υπόθεση συνεχίζεται. Έχουμε νέες έρευνες που έχουν να κάνουν με την εφορία. Αυτό το λέω. Αυτά τα τρία λοιπόν, offshore leaks, looks leaks και ε, Swiss Leaks, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα θέματα που δεν είναι διαρροές ε, leak, αλλά είναι ε, βάση δημοσίων στοιχείων και δεδομένων που είναι γνωστά, όπως η πρόσφατη έρευνα για την Παγκόσμια Τράπεζα. Στο μέλλον λοιπόν εμείς σε αυτό το όμιλος δημοσιογράφων θα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις και άλλες δημοσιεύσεις η οργάνωσή μας είναι μη κερδοσκοπική και δρεύει στην Ουάσιγκτον. Έχουμε 11 μόνιμους υπαλλήλους εκεί, αλλά πάνω από 190 δημοσιογράφους σε 65 χώρες που συνεργάζονται. Για να μάθετε ποια είναι τα θέματα που επιλέγουμε και βάζουμε όλη αυτή την ενέργειά μας. Έχουμε τρία κριτήρια για μια έρευνα για να ξεκινήσει. Μόνο αν το θέμα είναι παγκόσμιο και έχει παγκόσμια εμβέλεια και ενδιαφέρον. Δεύτερον, όταν είναι κάτι ε, συστηματικό, συστημικό και πρέπει να αποκαλυφθεί ένα σύστημα, όχι κάτι μεμονωμένο ή προσωπικές υποθέσεις. Και το τρίτο, αν μπορούμε εκ των προτέρων να εκτιμήσουμε ότι θα έχει πραγματικό αντίκτυπο αυτή η δημοσιογραφική έρευνα, όπως είναι ξεκάθαρο στην περίπτωση LuxLeaks. Λοιπόν, βεβαίως επίκυνται και νέες έρευνες. Τώρα πότε θα δημοσιευθούν και ποιο θα είναι το θέμα. Ε, θα σας αφήσουμε λίγο σε άγνωστα χαρτογράφητα είδατε. Ε, ο κ. Κλαστοντεύσκη λέει προηγουμένως ε, ρώτησε ε, τι κάνει η ερευνητική δημοσιογραφία και πώς πάει. Πολύ καλά. Ουδέποτε υπήρξε τέτοια διάσταση σε διασυνοριακή ερευνητική δημοσιογραφία, συνεργασία μεταξύ διαφορών δημοσιογράφων και οργανωμένων μάλιστα. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να πω ότι ε, ε, ε, χαίρει άκρας υγείας και εντός και εκτός της Ευρώπης. Ε, τις τρεις τελευταίες ε, μέρες είχαμε διάσκεψη στις Βρυξέλλες ερευνητικής δημοσιογραφίας περίπου 300 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο που ασχολούνται ε, με αυτό τον κλάδο της δημοσιογραφίας. Μπορεί να κάνει περισσότερη Ευρώπη, μπορεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ξέδωσε μια έκθεση όπου εκφράζει την εκτίμησή του για την ερευνητική δημοσιογραφία και τονίζει τη σημασία της. Ας πούμε στην καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει χρήματα για να υποστηρίξει την ερευνητική δημοσιογραφία που θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει ε, με διάφορους φορείς, ιδρύματα κτλ ή με υποτροφίες σε μεμονωμένους δημοσιογράφους. Υπάρχει πολύς χώρος εδώ για να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ασκούνται πιέσεις προς εμάς τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης των Λουξ Leaks και μετά, αν ασκήθηκαν τέτοιες πιέσεις ρωτήσατε, τα καλά νέα είναι ότι βάσει των άρθρων που δημοσιεύθηκαν παγκοσμίω, ούτε ο όμιλός μας, ούτε οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης ε, ε, που τα δημοσίευσαν ε, υπέστησαν διώξεις, ούτε μηνύσεις, ούτε τίποτα. Για τα άρθρα μιλώ τα ίδια. Δεν υπήρξε καμία νομική αμφισβήτηση και αυτό δείχνει και την ποιότητα της δουλειάς μας. Δεν αμφισβητήθηκαν τα δημοσιεύματα. Η κριτική ήταν από τις εταιρείες που θίγονται, που ισχυρίστηκαν ότι Είχαμε ε, ανακρίβειες, inaccuracies στα άρθρα, αλλά ποτέ δεν μας είπαν ότι αυτά που γράφεται είναι λάθος, ε, είναι ψευδή στοιχεία κτλ. Απειλές υπήρξαν ε, ότι θα μας μηνύσουν. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ο πρόεδρος μιας εταιρείας απείλησε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της εφημερίδας που το δημοσίευσε για συκοφαντική λέει δυσβήμιση, αλλά μετά καμία δίκη δεν ακολούθησε, ούτε μήνυσε. και ένα τελευταίο, λίγες μέρες πριν δημοσιευθούν τα Lux Leaks παγκοσμίω, που ήταν η 5η Νοεμβρίου του 2014, ο όμιλός μας έλαβε μία επιστολή από την Price Coopers τους δικηγόρους τους, που έλεγε ότι, και το παραθέτω στα αγγλικά, μία ασυνήθις ε, ε, δημοσίευση παρανόμως κτηθέντων στοιχείων μπορεί να έχει συνέχεια αστική ή ποινική για τους δημοσιογράφους. Αλλά αυτό είχε να κάνει με τη διαδικασία και όχι με το περιεχόμενο ε, των στοιχείων. Οι αντιδράσεις από τον υπόλοιπο κόσμο, πώς ε, έγιναν δεκτά αυτά τα LuxLeaks στην Ευρώπη και αλλού. Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι οργανώσεις. Για να προετοιμάσουμε την ακρόαση αυτή, δραστηριοποιήσαμε το δίκτυό μας και ζητήσαμε κάποια στοιχεία να μας δώσουν πρώτο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι ε, το Αμερικανικό κράτος δεν ανέβρασε καθόλου η κυβέρνηση. Αυτό είναι λίγο σαν ε, τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο που δεν βλέπει κανείς και δεν θέλει κανείς να αναφέρει. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Καμία αντίδραση από πλευράς αμερικανικής κυβέρνησης. Σε άλλες χώρες μπορώ να σας δώσω παραδείγματα, όχι όλα, στη Γερμανία ε, μια ομάδα εργασίας συστάθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και από τα Ομόσπονδα Κρατήδια και πρόσφατα βγήκε μια έκθεση ε, με αφορμή το LuxLeaks. Αποτέλεσμα δεν μπορούν ακριβώς να υπολογίσουν την οικονομική ζημία για τη Γερμανία. Είναι πολύ περίπλοκο, αλλά η ομάδα εργασίας λέει θα συνεχίσει την έρευνά της. Στην Ολλανδία Έγιναν ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο και η συζήτηση μετατοπίστηκε πολύ γρήγορα από το Λουξεμβούργο στην Ολλανδία, στην κατάσταση της κάτω χώρες που έχει και εκεί φορολογικά κίνητρα. Όπως γνωρίζετε, επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, κάλεσαν την Price Waterhouse Coopers ε, στη Βουλή και έβγαλα μια έκθεση πάρα πολύ επικριτική στην Σουηδία. Ο Υπουργός ε, Οικονομικών είπε ότι έχει έρθει η ώρα να αλλάξουν τα πράγματα στην Ευρώπη μετά το LuxLeaks όλα αυτά και επίσης είπε ότι οι σουηδικές πολυεθνικές θα πρέπει να έχουν πιο υπεύθυνη στάση στο μέλλον. Στη Φιλανδία έγινε συζήτηση στη Βουλή, στο Βέλγιο ακρόαση στη Βουλή όπου πήγαμε κι εμείς οι Βέλγοι δημοσιογράφοι του ομίλου αυτού και δώσαμε ε, ε, στοιχεία. Υπάρχει ε, ολόκληρη συζήτηση για το tax shift στη Δανία. Ήταν μαζικές οι αντιδράσεις. Ο υπουργό Οικονομικών και Φορολογίας ζήτησε έρευνα, διέταξε έρευνα για τα στοιχεία LuxLeaks, τα ντοκουμέντα που είναι και στην ιστοσελίδα μας. Και διεύρυνε και τον προπολογισμό που διαθέτει η Δανία σε αυτή την έρευνα. Και επίσης ε, η τοπική αυτοδιοίκηση στη Δανία δεν ε, μπορεί να προχωρήσει σε συμβάσεις με εταιρείες που χρησιμοποιούν φορολογικούς παραδείσους τους αποκλείουν από τους διαγωνισμούς. Ε, υπήρξαν και άλλες χώρες που δεν έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και στο Ισραήλ τώρα δεν έγινε καμιά τεράστια φασαρία. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το whistleblowing, τους καταγγέλλοντες, Α, να επαναλάβω λίγο. Ο διευθυντής μας, ο Gerald Trial, έχει ε, κάνει μια δήλωση ότι μία από τις φερόμενες ως πηγές ε, στο Λουξεμβούργο η στη ποινική δίωξη. Το διάβασα και στα αγγλικά ε, ε, η προστασία των πηγών και των καταγγελόντων είναι τόσο σημαντική για την κοινωνία όσο η ελευθεροτυπία. Οποιαδήποτε δίωξη δημοσιογράφων ή πηγών είναι επικίνδυνη και τονίζουμε τον θαραλέο και γενναίο ρόλο που παίζουν ε, μεμονωμένα πρόσωπα στην αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων. Ο ίδιος διευθυντής Gerald Ryle έκανε ε, και δήλωση ε, για τον κύριο Περά μετά τη δίωξή του και θέλω να σας τη διαβάσω σύντομα στα αγγλικά. Ο δημοσίευσε ε, τις της πρακτικές και αυτό ε, δημιούργησε μεγάλη συζήτηση καθώς επίσης και έρευνες για το LuxLeaks έπαιξε σημαντικό ρόλο, ε, αποκάλυψε στρατηγικές φοροαποφυγής από πλευράς του Λουξεμβούργου που είναι εις βάρος των κρατικών ταμείων και των ε, φορολογουμένων και ένα κράτος μέλος από τα ιδρυτικά της Ευρωπαϊκής ε, Κοινότητας δεν μπορεί να διώκει ε, έναν δημοσιογράφο κτλ. Αυτά ήταν οι επίσημες αντιδράσεις και του ομίλου μας των ερευνητικών δημοσιογράφων για την προστασία των καταγγελόντων και των δημοσιογράφων. Και με ρώτησαν επίσης αν υπάρξει διαφορά ανάμεσα στην προστασία των πηγών των δημοσιογράφων αφενός και την προστασία των καταγγελόντων αφετέρου. Βεβαίως υπάρχει διαφορά. Σε ό,τι αφορά την προστασία των πηγών, των δημοσιογράφων, το Βέλγιο έχει μια πάρα πολύ καλή νομοθεσία. Νομίζω ότι είναι υποδειγματικός ο νόμος παγκοσμίω για το πώς πρέπει να ρυθμίζονται αυτά τα πράγματα. Και αν χρειάζεστε έμπνευση, κοιτάξτε το βελγικό νόμο φτάνει μέχρι σημείου που όταν βελγικές μυστικές υπηρεσίες θέλουν να ερευνήσουν κάτι, ας πούμε το, τηλέφωνό μου να παρακολουθήσουν ή τον υπολογιστή μου, και μόνο το γεγονός ότι είμαι δημοσιογράφος χρειάζεται ιδιαίτερες εγγυήσεις. Δηλαδή η προστασία των πηγών είναι δεδομένη στο Βέλγιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένας καταγγέλων που θα έρθει να μου καταγγείλει κάτι θα έχει την ίδια προστασία. Δεν είναι πηγή. Ε, και μπορεί ξαφνικά να βρεθεί χωρίς εισόδημα γιατί τους απολύουν ε, τους καταγγέλλοντες. Δηλαδή ε, πάνε, καταγγέλουν, τους απολύουν και δεν βρίσκουν και ποτέ αλλού δουλειά. Αυτό είναι ένα ε, πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και δεν καλύπτεται από την προστασία των πηγών. Δηλαδή πρέπει να δοθεί απάντηση και στα δύο. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπρούξ, τελευταίος για πέντε λεπτά. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποια από τα ερωτήματα των μελών σας δείχνουν πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια και πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι οι κυβερνήσεις θα αλλάξουν το τι κάνουν με τη φορολογία θα βάλουν εντονότερο το στοιχείο της διαφάνειας. Ένα από τα θέματα που έδειξαν οι ευρωβουλευτές ήταν η νομιμότητα. Στις, ε, στα όσα έχουμε γράψει οι συνάδελφοί μου και εγώ επισημαίνει το γεγονός ότι οι δικηγόροι μας λένε ότι αυτά πράγματα είναι απόλυτα νόμιμα. Όμως όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι περιπτώσεις lax, LEAX, περιλαμβάνουν εταιρείε προσώψη στο Λουξεμβούργο, οι οποίες βεβαίως για να λειτουργήσει το σύστημα πρέπει να έχουν φορολογική έδρα στο Λουξεμβούργο. Γι' αυτό έχουν διάφορες προβλέψεις οι ε, διάφορες χώρε μέλη. Όμως υπάρχει και κάποια ουσία, υπάρχει δηλαδή και κάποια φορολογική ουσία. Αν δεν υπάρχει τότε είναι απόλυτα παράνομο. Γενικά. Άρα η υπόθεση ότι όλες οι υποθέσεις αυτές είναι απόλυτα νόμιμες δεν είναι αλήθεια. Τα τεστ που κάνουν οι φορολογικές αρχές ε, και εδώ είναι η μεγάλη σημασία της διαφάνειας και τα μίδια θα πρέπει να είναι αυτά που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Οι περισσότερες από τις ε, κυβερνήσεις των χωρών μελών όμως δεν είναι καν σε θέση να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Γιατί και οι φορολογικές τους υπηρεσίες δεν είναι επαρκώς τελεχωμένες, ειδικά σε περίοδους κρίσεων. Και δεν αμφισβητούν επαρκώς τα στοιχεία που τους δίνουν οι επιχειρήσεις. Ούτε μου φαίνεται ότι στο μέλλον ξαφνικά οι φορολογικές υπηρεσίες στις χώρες μέλη θα αρχίσουν να προσλαμβάνουν χιλιάδες φορολογικών επιθεωρητών. Επομένως τα αποτελέσματα αυτών των φορολογικών ε, συστημάτων εντός εισαγωγικών πρέπει να φωτιστούν έτσι ώστε τουλάχιστον να αναυποχρεούνται οι εταιρείε να εξηγούν με ποιον τρόπο πέτυχαν τα αποτελέσματα που πέτυχαν, δηλαδή να φορολογούνται σε τόσο χαμηλούς συντελεστές. Κάποιοι από τους βουλευτές μίλησαν και για τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ χωρών μελών για φορολογικές διευκολύνσεις. Τα αποτελέσματα γίνονται καθαρά όταν δείτε πού πληρώνουν τους φόρους τους οι επιχειρήσεις και με βάση ποιο κέρδος. Και αυτό, αυτή η υποβολή αναφορών ανά χώρα country by country reporting, είναι απόλυτα κρίσιμη. Και να δοθεί η δυνατότητα και στους αναλυτές και στους δημοσιογράφους να μπορούν να διερευνούν ποιες είναι ακριβώς οι δομές των επιχειρήσεων αυτών. Αυτές οι υποθέσεις Leaks που είναι εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, δεν ήταν παρά μόνο μια φωτογραφία ενσταντανέ που έδειξε μία εταιρεία λογιστών η οποία διερευνήθηκε τους τελευταίους μήνες ε, στο Ενωμένο Βασίλειο και έτσι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από το τι θεωρεί το κοινό και τι γίνεται πραγματικά. Και αυτά λοιπόν ξαναλέω ήταν υποθέσεις μιας λογιστικής εταιρείας για μια περίοδο 2-3 ετών και βεβαίω για μία μόνο χώρα που είναι το Λουξεμβούργο. Επαναλαμβάνω, επρόκειτο για φωτογραφία ενσταντανέ όλων αυτών των υποθέσεων. Ούτε μπορείτε να έχετε εξασφαλισμένου τους καταγγέλλοντε ότι δηλαδή κάθε τόσο θα βγαίνουν και θα καταγγέλουν για το τι έγινε. Και αν αυτά που λέει ο κ. Σπερά είναι σωστό, είναι σωστά, αυτοί αποτρέπονται κιόλα. Έχουμε και στο άλλο που ήθελα να πω τώρα πολλοί μιλούν για την προστασία των καταγγελόντων. Όση προστασία και να προσφέρεται όμως ένα καταγγέλλοντα, μπορεί να καταστρέψει τη σταδιοδρομία του. Χάνει τη δουλειά του και καταλήγει να μην έχει απολύτως τίποτα. Θα βρείτε ανθρώπους, καταγγέλλοντες δηλαδή, που όση η νομική προστασία και να τους προσφερθεί, η ζωή τους είναι κατεστραμμένη. Χρειάζεται λοιπόν και ανταμοιβέ στις ΗΠΑ προβλέπονται σημαντικότατες οικονομικές ανταμοιβέ. Ορισμένοι και ε, τη τάξη των εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων γιατί πήγε και στη φυλακή βέβαια αλλά τουλάχιστον πήρε και μια ανταμοιβή. Αυτή είναι και η τελευταία σκέψη που σας υποβάλλω. Ότι χρειάζεται δηλαδή και να προβλέψετε ανταμοιβέ για τους καταγγέλλοντες. Κουνάς, ένα λεπτό. Ναι, πολύ γρήγορα. Για να μην τα επαναλάβω όλα. Κάτι που δεν ε, διευκρινίστηκε για την αυτόματη ανταλλαγή των ε, συμφωνιών. Αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη, εφόσον υποτίθεται ότι είχε προβλεφθεί, ε, καλή την πίστη να μεταφέρουν τις πληροφορίες για τις συμφωνίες τους και σε άλλες όλες αρχές. Διοικητικώς έτσι οι αρχές ε, θα έπρεπε να είναι εξοπλισμένες βέβαια για να μπορούν να αντιμετωπίσουν, να καλύψουν τα δεδομένα αυτά και αν οι συμφωνίες αυτές ήταν προσβάσιμες και στο ευρύ κοινό, τα πράγματα αυτά ήταν τέλεια, διότι νομίζω ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ξέρουν τι μεταχείριση επιφυλάσσεται σε επιχειρήσεις στη χώρα τους. Και για, την, ε, για τον αθέμητο ανταγωνισμό που πολλές φορές έχει αναφερθεί εδώ στην ε, Επιτροπή. Υπάρχουν ε, επιχειρήσεις που είχαν ευνοϊκής μεταχείρισης από τη μια και από την άλλη οι υπόλοιπε μπορεί να μην το γνωρίζουν. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουν πρόσβαση από τέτοιες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω όλους ε, τους όλα τα μέλη του Consortium για την ακρίβεια των απαντήσεών τους και για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα θα ε, συμπεράνουμε μεταξύ άλλων και όπως ισχύει και για τους περισσότερους που ακούσαμε εδώ ως μάρτυρες, τους δύο τον κύριο Τόιρερ και την κυρία Φερέιρα, μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας για να εμπαθύνουν σε μερικά πράγματα. Έχω ε, να σχολιάσω για το Γιβραλτάρ, ε, γιατί από θα περάσουμε από το Λουξεμβούργο, το Γιβραλτάρ, μετά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιούνιο, 18 έκτου, Και βεβαίω εκεί θα δούμε και τι αντιδράσει τη Μαδρίτη. Αλλά έχετε κάνει, υπάρχουν υπάρξει δημοσιεύματα σε πολλά μέσα των κρατών μελών για το Λουξ Leaks. Και εσεί έχετε κάνει πολλέ δημοσίευσει. Θα ήταν καλό λοιπόν να μπορείτε να μα δώσετε τον πλήρη κατάλογο για να συμπληρώσουμε ε, το σώμα των πληροφοριών που διαθέτουμε και να μα πείτε κατά πόσον είχατε τη μια ή την άλλη συνομιλία με κάποια εθνική φορολογική αρχή. Επίσης, όπως περιγράψατε τις ευθύνε και τις αρμοδιότητες των ερευνητών δημοσιογράφων, Κάποιος από εσά είπε ότι θα έπρεπε να υπάρχει οικονομική βοήθεια από, μια, ε, από κάποια πηγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όπω και αν είναι αυτή η μορφή από ίδρυμα, αλλά διαφωνώ. Stop. Διότι όποιο μιλάει για κρατική παρέμβαση εννοεί και πάυση τη ελευθερωτυπίας αναστολή τη ελευθερωτυπίας της ελευθερίας έκφρασης ε, μην ξεχνάμε και την έκφραση που μπορεί να τη λέω με κακή προφορά στα λατινικά, ε, φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντες. Δηλαδή, ε, στους δημοσιογράφους έχω να πω προσοχή, προσοχή στο κράτος σε περίπτωση που σας δίνει ακόμη και τα ωραίτερα δώρα, ο καθένας στο ρόλο του. Νομίζω ότι πολύ καλά καταλάβατε, το υπενηθήκατε πολύ από εσάς ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, ε, εάν αυτά που ανακαλύψατε ήταν ε, νόμιμα ή παράνομα. Το δύσκολο πρόβλημα δεν είναι να καλυφθεί αυτό που δεν είναι νόμιμο. Η μεγάλη δυσκολία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά πρέπει να λάβει μέτρα εφόσον πρόκειται για κάτι παράνομο, είναι ότι υπάρχει η φόρα που φυγεί, διότι υπάρχουν 28 διαφορετικά συστήματα. Είναι εφικτό και γίνεται διαρκώς, ιδίως για όλες τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν συμβουλές από ε, εταιρείε συμβούλων, consulting που έχουν ε, μεγάλες γνώσεις, ε, να διαφεύγουν από τι φορολογικές αρχές ενό κράτου μέλου. διότι κάπου μια δαπάνη θεωρείται ως ε, οικονομική ε, συναλλαγή που εκπίπτει του φόρου από μια χώρα, ενώ μια γειτονική χώρα μπορεί να το θεωρεί μέρισμα που εκπίπτει στην συγκεκριμένη αυτή χώρα, αλλά όχι στην προηγούμενη. Εδώ μιλάμε για δάνεια ευρύδια ή για μέτρα ευρύδια, κάτι που υπόθηκε προηγουμένως. Άρα, με άλλα λόγια, όταν ε, ανήκει κανείς σε μια οικονομική οικογένεια, μια οικογένεια λαών, μια ε, οικογένεια πολιτισμών και νοοτροπιών με κοινέ αξίε όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ορισμένου τομεί, το γεγονό ότι υπάρχουν διαφορετικοί κανόνε οδηγεί σε καταστάσει άδικε και ανήθικε. Σε ορισμένου τομεί. Δεν λέω παντού. Υπάρχει κατανομή αρμοδιοτήτων, υπάρχει επικουρικότητα και το καταξής. Όμως εδώ βρισκόμαστε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, ένας από τους δρόμους που πρέπει να εξερευνήσουμε, κάτι που άρχισε να συζητιέται ήδη πριν από χρόνια, είναι να καταφέρουμε να ορίσουμε με τρόπο κοινό τη φορολογική βάση για τα κέρδη των εταιριών. Εάν είχαμε έναν και μόνο κανόνα αντί για 28, δεν θα είχαμε πλέον τόσες πολλές περιπτώσεις και ευκαιρίες να φοροαποφύγει κανείς. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο τρομακτικό πρόβλημα. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η βάση, πώ θα καταναμηθεί μεταξύ των κρατών. Αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση ε, δρά και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό κράτη. Υπάρχουν ομοσπονδιακά κράτη που το χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα, τη γνωρίζει τη κοινή φορολογική βάση όσα. αλλά το θέμα είναι πώ θα εφαρμοστεί. Ιδίω με την ψηφιακή οικονομία που δεν προλάβαμε να την αναπτύξουμε σήμερα το απόγευμα, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Αυτό είναι ένα θέμα επί του οποίου θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά. Και για το οποίο οι μαρτυρίες, οι συμβουλές, οι συστάσεις των ε, δημοσιογράφων που έχουν ειδικέ γνώσει θα μας ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες. Σας ευχαριστώ, ε, σας απελευθερώνω. Διακόπτω για δύο λεπτά την συνεδρίαση για να φύγετε από την αίθουσα και μετά θα συνεχίσουμε με το επόμενο πάνελ.

ξαναρχίζει η συνεδρίαση. Παρακαλώ καθίστε και ησυχάστε. Είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της μακράς ακρόασης και αφού ακούσαμε τις μαρτυρίες καταρχήν και κλεισμένων των θύρων των πληροφοριοδιώτων και μετά των δημοσιογράφων Αλλάζουμε τώρα λίγο προσέγγιση για να δούμε τις αναλύσεις και συστάσεις τριών εξεχόντων πανεπιστημιακών που ειδικεύονται σε θέματα επιχειρησιακής φορολογίας. Δομινίκ Μπερλέν. που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 2 ο Δόκτωρ Γκαβριέλ Τσούκμαν που είναι Assistant Professor στο London School of Economics και ο Δόκτωρ Χακίμ Αρίμ Αχίμ Ντάρφερ. Θα ζητήσω λοιπόν όπως και πριν πρώτα από τους εισηγητές να κάνουν μια εισήγηση και ο καθηγητής Μπερλέν είχα με πει ότι είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση που τον, υποχρεώνει, που τον αναγκάζει να φύγει σε λίγο και άρα αν μπορούν τα πρώτα ερωτήματα να απευθυνθούν σε εκείνον θα μας είναι ευγνώμων. και κατά τα άλλα θα συνεχίσουμε γραπτός, ηλεκτρονικά κτλ. Ελίζα, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα από τα θέματα που θα ήθελα να θίξω είναι πώς θα ποσοτικοποιήσουμε αυτά που λέμε. Θα έχετε φαντάζομαι όλοι κάποιους υπολογισμούς, κάποια επιχειρήματα, κάποιες εξηγήσει μέχρι που μπορούμε να πάμε για να αντιμετωπίσουμε τα spillover effects από μια χώρα σε μια άλλη, μέσα στην Ευρώπη ιδίω. Δεύτερον, πολύ σημαντικό αλλά γνωρίζουμε πολύ λίγα γι' αυτό είναι η φορολογική παράδειση και τα ειδικά νομικά καθεστώτα που τους αφορούν. Υπάρχουν ειδικέ δικαιοδοσίες νομικές μέσα στην Ευρώπη αλλά με ειδικό καθεστώς εκτός Ευρώπης ή, ή απικίες της ε, Βρετανικής, ε, του Βρετανικού στέματος κτλ. Μέχρι πού μπορούμε να πάμε λοιπόν από ευρωπαϊκής απόψεως, τι μπορούμε να κάνουμε και τι να, δεν μπορούμε να κάνουμε. Τρίτον, ένα ερώτημα που συχνά θέτω στον εαυτό μου. Εσείς που τα έχετε επεξεργαστεί αυτά τα στοιχεία Πώς εξηγείτε το ότι πολλές χώρες μέλη που χάνουν μεγάλα ποσά φορολογικών εσόδων πηγαίνουν στο Συμβούλιο και δεν θέτουν το θέμα. Γιατί. Είναι αλήθεια ότι όλοι παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Είναι των ίδιων διαστάσεων. Μιλήσαμε για το Λουξεμβούργο αλλά Υπάρχουν βέβαια οι συνήθεις ύποπτοι, αλλά εκτός αυτών, γιατί δεν παραπονείται κανείς, ποιος είναι ο λόγος. Και τέλος, η διαφορά μεταξύ του νόμιμου, αλλά που στρεβλώνει την αγορά, και του παράνομου, όταν γίνονται οι υπολογισμοί των φορολογικών αυτών απολειών λόγω τέτοιας φορολογικής πρακτικής. Ευχαριστούμε Ελίζα. Μιχαήλ το Γιωράρκ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο δόκτωρ Τούτμαν και ο δόκτωρ Τότμαν είναι άνθρωποι που τους πρότεινα εγώ και γι' αυτό Χαίρομαι, Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκονται εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουν πάρα πολλές δημοσιεύσεις. Το θέμα είναι να γίνει μια εκτίμηση των διαστάσεων του φαινομένου της φοροαποφυγής ή φοροαποφυγής και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να γνωρίζω πού βασιστήκατε για αυτές τις εκτιμήσεις. Ακούγονται νούμερα που, φτιάχνουν, που που φτανουν το 1-3 εκατομμύριο ετησίως που χάνεται από φορολογικά έσοδα. Μιλάμε για τεράστια νούμερα. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε σε ποια δεδομένα βασιστήκατε. Το δεύτερο ερώτημα. Στις ε, έρευνές σας ε, γίνεται σαφές πως πρόκειται για ένα σύστημα. Μιλάτε για μια βιομηχανία φοροαποφυγής τα λέω τώρα αυτά από μνήμης, αυτά που έχετε γράψει. Δηλαδή πρόκειται για μια σειρά επιχειρήσεων που δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να βελτιστοποιούν ε, τους φόρους ή να αποφεύγουν τους ε, φόρους ή να φτάνουν μέχρι και την παρανομία, την φοροδιαφυγή. Ε, επιμένετε σε αυτά τα οποία είπατε και ε, ποια είναι, ποιοι είναι εδώ πέρα οι κύριοι δράστες. Και τρίτον, μιλάτε για λύσεις, κάνετε κάποιες προτάσεις για το τι μπορούν να κάνουν τα εμπλεκόμενα κράτη και ο Εδώ πέρα μιλάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια κοινή φορολογική εταιρική βάση. Έχουμε επίσης ε, τις ε, προτάσεις ε, για καλύτερες φορολογικές έρευνες μέσω κοινών ελέγχων, επιτόπιων ελέγχων. Συζητάμε την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Κατά την άποψή σας υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα έπρεπε να λάβουμε. Ή θεωρείτε αυτά τα οποία προτείνουμε που βασίζονται στους κανόνες του ΩΣΑ ότι επαρκούν. Και τέλος Εμεί επικεντρωνόμαστε στα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης. Τώρα όμως βλέπουμε ότι γρήγορα γρήγορα ακούγονται και άλλες χώρες. Ε, τα νησιά της Μάχης, Τζέρσι και Γκένσι, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή τα νησιά της Καραβικής, ε, Βερμούδες, ε, Μπαχάμες, Παρθένες νήσι, Βανουάτου, στον Ειρηνικό, Πρέπει να κανείς να ψάξει την υδρόγειο. Αυτή η παγκόσμια διάσταση λοιπόν μπορεί να αγνοηθεί ή πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ τους τρεις ομιλητές μας. Καταρχάς, για τα έγγραφα που μας έστειλαν, όχι όλοι, αλλά κάποιοι, και για τα προφορικά τους ε, σχόλια που θα κάνουν τώρα. 7 λεπτά ο καθένας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο μετά στους εκπροσώπους ε, των πολιτικών ομάδων και μετά να δοθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις. Ο καθηγητής Μπερλάν. Από όλα όσα άκουσα πριν, ε, άσε να σκέφτομαι, έχω θέση σε αυτή τη συζήτηση. Άκουσα πολύ να γίνεται λόγος για διοντολογία για υπεύθυνη συμπεριφορά, για ανήθικη συμπεριφορά. Εάν ε, έχω κάποια πραγματογνωμοσύνη, αυτή δεν είναι η διοντολογία, δεν είναι τα ηθικά θέματα, αυτό το αφήνω στους πολιτικούς, γιατί αυτοί θα πρέπει να δώσουν λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα μιλήσω για τα νομικά θέματα. Εκεί θα περιοριστώ, γιατί αυτό είναι ο τομέα τη ε, εμπειρογνωμοσύνη μου και γι' αυτό είμαι εδώ παρόν. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις και θα αφήσω το λόγο στους ε, βουλευτές να κάνουν ερωτήσεις. Ε, με ρωτήσατε αν, έχετε, αν έχω προτάσεις ή λύσεις. Έχω κάποιες ιδέες, αλλά η πρώτη μου ιδέα είναι να πούμε σε αυτήν την Επιτροπή να είναι πάρα πολύ συνετή και προσεκτική, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος να ανακατευτούν, να κατέψει πολλά προβλήματα που είναι διαφορετικής προέλευσης. Πολύ σωστά δείξατε στο τέλος της πρώτης συνεδρίασης. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν παράνομα, παράνομες συμπεριφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε όλα τα εργαλεία για να τα καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα, αυτές τις συμπεριφορές. Το πρόβλημα δεν είναι η παρανομία κάποιων συμπεριφορών. Φυσικά θα πρέπει να τις καταπολεμήσουμε. Ε, και έχουμε τα μέσα για να το κάνουμε. Το θέμα που θέτει η Επιτροπή σας είναι τι κάνουμε έναντι συμπεριφορών που κατά κανόνα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι νόμιμες συμπεριφορές. Και εκεί μπαίνει το θέμα της διοντολογίας. Ε, και των προβληματικών πολιτικών. Γιατί, όπως είδαμε, κάποιοι από τους προλαλήσαντες ε, εκπλήσονταν που δεν αντιδρούμε απέναντι σε κάποιες νόμιμες συμπεριφορές. Μα πώς να αντιδράσουμε όταν πρόκειται για μια νόμιμη συμπεριφορά. Και αν είναι νόμιμη συμπεριφορά, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία προσφυγή νομικής φύσεως, αν η συμπεριφορά είναι απόλυτα νόμιμη. Εάν είναι αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε και αν βρίσκουμε σοκαριστικές μερικέ ε, νόμιμε συμπεριφορέ, θα πρέπει να αλλάξουμε του κανόνε. Ο στόχο, λοιπόν και ο λόγο ύπαρξη τη Επιτροπή είναι να προτείνει λύσει για να αλλάξουμε το δίκαιο, ούτω ώστε να εξαφανιστούν αυτέ οι συμπεριφορέ, οι οποίε είναι ασύμβατε με την ε, δεοντολογία, την ηθική κτλ. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξεκινήσω από αυτό. Ήθελα να το πω αυτό γιατί νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνο για την Επιτροπή να θέλει να κάνει πάρα πολλά και να χάσει την αξιοπιστία της ε, λόγω του τεράστιου εύρου των προτάσεων που θα κάνει. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι δεν σημαίνουν τα ίδια πράγματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι πρόβλημα αυτό. Το, το tax ruling, ας πούμε. Το ίδιο, το βασικό σας θέμα. Ε, στα γαλλικά λέγεται rescrit φορολογικές συμφωνίες. Δεν είναι ίσως καλή μετάφραση του αγγλικού tax rulings. Αν πάρουμε ένα παράδειγμα του τι εννοείται στο Λουξεμβούργο tax ruling, είναι αυτό που λέμε στη Γαλλία εγκρίσει, agrément, Συμφωνίε. Δηλαδή, οι φορολογικέ διοικησει ε, μεταχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο, με εξατομικευμένο αν θέλετε τρόπο, μια συγκεκριμένη ε, επιχείρηση. Ε, στρεβλώνοντας λιγάκι την ε, νομοθεσία στα πλαίσια του γενικού συμφέροντος. Ενώ το ΕΣΚΡΙ, και σας έδωσα προηγουμένως ε, ποια είναι τα άρθρα του, του κώδικα, είναι κάτι άλλο, στη Γαλλία τουλάχιστον, έτσι. Έχετε την επιλογή να ερμηνεύσετε, να ερμηνεύσει δηλαδή η εφορία το γενικό νόμο, γιατί το ζητάει μια επιχείρηση, έτσι, γιατί δεν κατάλαβε καλά, γιατί ο νόμος δεν είναι σαφής. Ή η εφορία επιβεβαιώνει τροποντινά σε μια επιχείρηση ότι λαμβάνοντα υπόψη τη δραστηριότητά τη, αυτή η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη θα εφαρμοστεί. Και το όφελος είναι ότι μπορεί να αντιτάξει αυτό το, αυτή τη συμφωνία, ας πούμε, ε, απέναντι στη διοίκηση και η διοίκηση δεν μπορεί εκ των υστέρων να έρθει, ας πούμε, αναδρομικά, ας πούμε, και να δώσει μια άλλη ερμηνεία Τη δόθηκε αυτή η ερμηνεία τη επιχείρηση, τη χρησιμοποιεί λοιπόν αυτή την ερμηνεία. Επομένω, θα πρέπει νομικώ πώ να πλαισιώσουμε σωστά το πρόβλημα για να δώσουμε και την κατάλληλη λύση. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί και θα επανέλθω αφού δώσω το λόγο και στου άλλου ομιλητέ. Πολύ ωραία κύριε καθηγητά. Στη Γαλλία λοιπόν υπάρχουν 3.000 τέτοια ρεσκρή κάθε χρόνο. Και κάτι ανάλογο γίνεται σε όλες τις χώρες. Και δεν είναι κάτι καταδικαστέο, είναι και χρήσιμο. Δίνει τη βεβαιότητα στον χρήστη για το τι δικαιώματα έχει. Μάλιστα πολλές φορές οι σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το ζητούν. Πάμε τώρα στον μεσαίο μιλητή. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που με δέχεστε σήμερα. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα ζήτημα που προέκυψε αρκετές φορές στη συζήτηση. Υπό το φως των όσων μάθαμε από τα LuxLeaks τι μπορεί να γίνει για την εταιρική φοροαποφυγή, πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί το σύστημα αυτό το οποίο λέω είναι πως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης των πολυεθνικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λειτουργεί πλέον το σύστημα των 28 διαφορετικών εταιρικών φορολογικών συντελεστών με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του κέρδους. Και βεβαίω είναι ένα ζήτημα που πάει πέρα από την Ένωση, δηλαδή το πώς φορολογούν τις ε, εταιρείε αυτές και εκτός της Ένωσης είναι προβληματικό. Αλλά δεν περιορίζεται εντό τη Ένωση. Κοιτάξτε, ο τρόπο αυτό τη φορολογία εφευρέθηκε το 1920, πριν από έναν αιώνα, όταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο είχαμε την εταιρική φορολογία και στη δεκαετία του 1920 η κοινωνία των εθνών ανησύχησε πως πολλές χώρες θα προσπαθούσαν να φορολογήσουν το ίδιο ευρώ κέρδους ε, δύο φορές και θα είχαμε διπλή φορολογία. Για να αποφευχθεί η διπλή φορολογία, η κοινωνία των εθνών ζήτησε από τέσσερις οικονομολόγους να σχεδιάσουν κάποιους κανόνες για να φορολογήσουν τις πολυεθνικές και να μην υπάρχει διπλή φορολογία. Ο βασικός κανόνας που ισχύει μέχρι και σήμερα είναι αυτό το οποίο λέμε ενδομιλικές ε, συναλλαγές που είναι ο βασικός πυλώνας ε, των ε, φορολόγησης των επιχειρήσεων. Δηλαδή, ας πάρουμε μια γερμανική εταιρεία η οποία πουλάει καφέ, έχει μια βραζιλιανική φυγατρική. Εκεί πέρα παράγεται ο καφές ε, και η νητρική εταιρεία στη Γερμανία κάνει εισαγωγή από τη Βραζιλία και ε, τον διανέμει στους ε, Γερμανούς καταναλωτές. Αν δούμε ολόκληρο τον όμιλο, μέρος των κερδών δημιουργήθηκε στη Βραζιλία και μέρος των κερδών δημιουργήθηκε με τη διανομή και την πώληση καφέ στην ε, Γερμανία. Πώς καθορίζουμε λοιπόν πού ακριβώς δημιουργήθηκε το κέρδος. Έχουμε λοιπόν αυτές τις ενομιλικές συναλλαγές και υποθέτουμε ότι οι δύο αυτές εταιρείε, η θηγατρική και η μητρική, είναι τελείως ανεξάρτητες η μία από την άλλη και εμπορεύονται μεταξύ τους ε, σαν να μην είχαν καμία σχέση. Οπότε η γερμανική εταιρεία θα κάνει εισαγωγή καφέ από την βραζιλιάνικη θηγατρική της στην τιμή της αγοράς. Και αυτό τελικά θα δημιουργήσει κάποιο κέρδος φορολογητέο στη Βραζιλία και κάποιο κέρδος φορολογητέο στη Γερμανία. Αυτές είναι οι ενδομιλικές συναλλαγές πολύ απλά δεν λειτουργεί το σύστημα πλέον για δύο λόγους. Το ένα είναι πως ε, είναι αδύνατο να παρακολουθήσουμε τα δισεκατομμύρια αυτών των ενδομηλικών συναλλαγών ε, που λαμβάνουν χώρο κάθε χρόνο. Δεν μπορούν να το κάνουν οι φορολογικές αρχές, ειδικά σε ένα πλαίσιο λιτότητας, χωρίς ε, πόρους. Και το δεύτερο είναι πως σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποια τιμή αναφοράς αγοράς για τις ενδομιλικές συναλλαγές. Δηλαδή ποια είναι η τιμή, ποια είναι η αξία του σήματος ε, της Apple ε, ή της Microsoft, ε, άιλου, κεφαλαίου, ποια είναι η αξία ενός αλγόριθμου. Δεν υπάρχει συναλλαγή με τρίτα μέρη, οπότε δεν μπορεί να υπολογιστεί η αξία κάποιων πραγμάτων. Και εκεί πέρα ακριβώς έχουμε τις φορολογικές αποφάσει. Δηλαδή δεν υπάρχει τιμή αναφοράς, οπότε συμφωνήσουμε να ορίσουμε μία τιμή για αυτή την ε, συναλλαγή. Και σε πολλές περιπτώσεις όπως τα LuxLeaks η τιμή η οποία καθορίζεται είναι τέτοια ώστε το κέρδος σε τελική ανάλυση φαίνεται ότι γίνεται στη χώρα με τη χαμηλότερη φορολογία όπως τη Βερμούδα που είναι 0% η εταιρική φορολογία και οι ζημιές γίνονται στις μεγάλες οικονομίες, στη Γερμανία ή τη ΣΥΠΑ κτλ. Οπότε, κατά μία έννοια, το πρόβλημα δεν είναι οι αποφάσεις αυτές. Ε, οι αποφάσεις αυτές Απλά είναι μια ενσάρκωση, μια εκδήλωση του παράλογου αυτού συστήματος. Δηλαδή μπορούν οι εταιρείε να φανούν ότι τα κέρδη τους γίνονται στις χώρες με τη χαμηλή φορολογία. Υπάρχει κάποια βεβαιότητα; γιατί μπορεί να ισχύει αυτό σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις και λένε οι φορολογικές αρχές ότι θα απομακρύνουμε έτσι αυτή την αμεβαιότητα. Χωρίς αυτό ο κίνδυνος είναι ότι θα πληρώσει μια εταιρεία 1, 2, 3 πραγματικό εταιρικό φόρο. Ενώ με τις αποφάσεις αυτές θα πληρώσει 1% σίγουρα. Αυτό είναι το νόημα. Ποια είναι η εναλλακτική λοιπόν. Η εναλλακτική είναι να εγκαταλειφθεί αυτή η φαντασίωση ότι είναι ανεξάρτητες οι θηγατρικές και να μιλήσουμε για ενοποιημένη φορολογία. Μιλάμε για τα ενοποιημένα κέρδη της Microsoft, ας πούμε, τα παγκόσμια ενοποιημένα κέρδη μιας εταιρείας σαν τη Microsoft και μετά τα κατανέμουμε αναχώρα με βάση μια κλίδα κατανομής. Είναι δύσκολο να σχεδιαστεί αυτό. Όχι είναι ένας απλός κανόνας, είναι οι πωλήσει. Κατανέμουμε το κέρδος με βάση το που γίνονται οι πωλήσει. Π.χ. εάν 10% των πωλήσεων γίνεται στη Γερμανία, 10% των παγκόσμιων ενοποιημένων κερδών είναι φορολογητέα στη Γερμανία. Εντάξει, μπορεί να γίνει αυτό εντός της Ένωσης πάρα πολύ απλά για εταιρείες που λειτουργούν στις 28 χώρες. Αυτό κάνουν οι ΕΠΑ για τον πολιτιακό φόρο πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν οι πολιτείες γιατί δεν είναι σαν τα κράτη της ε, Ένωσης συνειδητοποίησαν πριν από δεκαετίες ότι θα είναι αδύνατον και εφαρμόζουν αυτό το σύστημα της κατανομής. Οπότε ας το κάνουμε στην Ευρώπη. Μπορούμε Εκεί πέρα, αυτό είναι το νόημα νομίζω της ε, κοινή ε, εταιρικής φορολογικής βάσης. Το συζητάμε εδώ και χρόνια, δεκαετίες. Τι περιμένουμε. Η μόνη λογική πολιτική αντίδραση στο LuxLeaks είναι να καταλήξουμε επιτέλους σε μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, σαφέστατο. Και τώρα ο κύριος Ακίμ Ντάρφερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω μερικά λόγια σαν εισαγωγή και μετά θα απαντήσω σε ερωτήσεις που τέθηκαν. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε το πλήρες εύρος του προβλήματος δεν έχουμε αξιόλογα στοιχεία, αξιόπιστα στοιχεία για τα ποσά για τα οποία μιλάμε. Δύο παραδείγματα. Η ελβετική κυβέρνηση μας είπε ότι 800 εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν φορολογηθεί στην ελληνικών χρημάτων δεν έχουν φορολογηθεί. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ψέμα. Ο Ότερ που ήταν παρόν πριν είχε πλήρη στοιχεία της τράπεζας Julius Fair που έχει μερίδες στην αγορά περίπου 3% και μου είπε ότι και μόνο αυτή η τράπεζα είχε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ελληνικών χρημάτων. Επομένως δεν είναι αληθή τα συνολικά ποσά. 80 μάλλον δισεκατομμύρια είναι το συνολικό ποσό ελληνικών χρημάτων στην Ελβετία και αυτό το διάβασα και από άλλη πηγή. Δεν είναι αξιόπιστα λοιπόν τα στοιχεία. Δεύτερο παράδειγμα. Η Ελβετία μας είπε ότι έχει μια στρατηγική σύμφωνα με την οποία στην Ελβετία δεν υπάρχουν πια παράνομα χρήματα. Ούτε αυτό το πιστεύω. Από τα στοιχεία που έχω από την τράπεζα αυτή την ίδια Γιούλιου Fair θα υπολόγιζα περίπου 10% χαμηλότερα τα γερμανικά χρήματα από φοροδιαφυγή στην Ελβετία. Λιγότερο από 10% από τα χρήματα αυτά έχουν επιστρέψει στη χώρα. και αυτό συμφωνεί και με αυτό που μας είπε πριν από τέσσερα χρόνια ο πρόεδρος αυτής της τράπεζας είπε όλα αυτά τα κόλπα από τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσουν σε 25% περισσότερων γερμανικών χρημάτων να φεύγουν από την τράπεζά μας, όχι παραπάνω. Δεν ξέρουμε λοιπόν τα ακριβή στοιχεία, ούτε πριν ούτε μετά η Ελβετία και οι Ελβετικές τράπεζες μας λένε ότι άλλαξαν τα πράγματα, ότι... Αλλά μόνο ένα γενικό εύρος μπορούμε, α, το γενικό εύρος μπορούμε να το υπολογίσουμε μόνο αν ξέρουμε τι υπήρχε ακριβώς πριν την αλλαγή. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Τα στοιχεία από το LuxLeaks και το SwissLeaks να αναφερθούν και με ονόματα να διατεθούν για τους ερευνητές να είναι πραγματικά στοιχεία. Δεύτερον, να μην ξεχνάμε ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι γενικά καλό πράγμα, αλλά πρέπει να είναι διαφανής. Και δεν βλέπω γιατί πρέπει να πούμε αν είναι νόμιμο ή παράνομο από τη μία ή αν είναι ηθικό ή ανήθικο από την άλλη. Υπάρχει και κάτι ενδιάμεσο. Ο ανταγωνισμός λοιπόν πρέπει να είναι διαφανής και να υπόκειται σε όλα τα νόμιμα μέσα ελέγχου που έχει στη διάθεσή της μια πεπολιτισμένη κοινωνία. ο δημοκρατικός έλεγχος υπάρχει και έπειτα ανοιχτή και διαφανής αγορά και τρίτον δικαστικός έλεγχος και τα τρία αυτά στοιχεία έχουν παραβιαστεί σε αυτές τις ειδικέ συμφωνίες στο Λουξεμβούργο. Δεν είναι ηθικό λοιπόν θέμα, είναι θέμα παραβίασης ορισμένων βασικών αρχών που συνιστούν την ένωση, ένωμη τάξη, δημοκρατία κλπ. Και αυτές οι ειδικέ συμβάσεις χωρίς κανέναν κοινοβουλευτικό έλεγχο ούτε καμία ευκαιρία ενός ανταγωνιστή να τον μηνύσει για στρέβλωση του ανταγωνισμού και χωρίς καμία διαφάνεια ή δυνατότητα άλλων χωρών να ανταγωνιστούν με κίνην. Να επιμείνουμε λοιπόν στις αρχές αυτές. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για ηθική, απλώς να τηρηθούν οι αρχές. Κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ότι εγώ δέχομαι τη συμμόρφωση με μέτρα δίωξης αλλά υπάρχει πολύ και πολύτιμη έρευνα για τη συμμόρφωση, παράδειγμα. Συμμόρφ, φορολογική συμμόρφωση είναι υψηλότερη όταν η φορολόγηση γίνεται τοπικά. Πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο πώς εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Όταν πληρώνει κανείς φόρους τοπικά γνωρίζει κανείς γιατί και σε ποιον πληρώνει. Υπάρχει υψηλότερη συμμόρφωση λοιπόν και δεν χρειάζονται μέτρα δίωξης τα οποία θα έπρεπε να είναι μόνο το τελευταίο μέτρο που θα έπρεπε να λάβουμε αν δεν γίνεται αλλιώς. Και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι επειδή η πιθανότητα σύλληψης των φοροδιαφευγόντων στη Γερμανία είναι μόνο 10% τα μέτρα δίωξης δεν δουλεύουν ή δεν δουλεύουν αρκετά. Χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Επίσης ήδη τονίστηκε ότι ο ρόλος των, πληφορο, των πληροφοριοδοτών Μιλήσαμε ήδη για τις συνέπειες που είχε ο νόμος Dodd-Frank στις Ηνωμένε Πολιτείε 25 με 30% του προστίμου που είχε επιβληθεί στην εταιρεία ε, το κατέδωσε αυτός ο άνθρωπος αυτή η γκρίζα περιοχή που υπάρχει δεν είναι κάτι πολύ ωραίο. Τέλος, θα χρειαζόταν μια συντονισμένη προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένα μόνιμο δίκτυο think tank σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις συνεχείς αλλαγές της πολιτικής που ισχύει για τη φορολογία καθώς και τον πολλαπλασιασμό των μέσων για φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια και σας ευχαριστώ μια δεύτερη φορά για το ότι τηρήσατε το χρόνο. Από το ΕΛΚ, ο κύριος Τόμ Βάντεν Κάντελαρ. Από το ΕΛΚΑ. Ο τελευταίο ομιλητή ουσιαστικά με κάλυψε, αλλά θέλω να μου απαντηθεί και το εξή. Πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνουν ε, μέτρα για να αντιμετωπίσουν ε, τι καταχρηστικέ φορολογικέ συμφωνίε ή φορολογικέ πρακτικές και υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μια παγκόσμια λύση στο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ακούσουμε μια σειρά από από ευρωβουλευτέ, από τους σοσιαλιστές τώρα, η κυρία Περβάνς Μπερές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο σειρές ε, les Πρώτον, τα μέσα που έχουμε για να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Ο πρώτος μας προσκεκτημένος είπε πολύ σωστά ότι ο στόχος της Επιτροπής μας είναι να επικεντρωθεί στο θέμα των ruling, των συμφωνιών, δηλαδή των φορολογικών συμφωνιών. Οι φορολογικές συμφωνίες, τα ruling, είναι ένα σύνολο. Εμείς μπορούμε να αυτοπεριοριστούμε, αλλά βλέπουμε και από τις παρεμβάσεις σας ότι κάτι ξεφεύγει. Και εκεί βλέπουμε ότι το θέμα της διαφάνειας, ε, της συμπεριφοράς των ανθρώπων είναι σημαντικό σε αυτές τις ιστορίες. Γιατί το ruling η βελτιστοποίηση, η φοροδιαφυγή τρέφεται από τη μυστικότητα και μας επιτρέπει να εξαπατήσουμε απέναντι στα άλλα κρατημέλη, απέναντι σε άλλες εταιρείες. Κύριε Ζούκμαν, σε σας απευθύνομαι γιατί ε, στα γραπτά σας μιλάτε για ένα είδος αρχείου, παγκόσμιου, όπου θα έχουμε μία απεικόνηση πολύ σαφή του τι συμβαίνει. το G20 του Ιουνίου του 2012 νομίζω ότι σημειώθηκε πρόοδος. Έγινε μία αρχή για το Διοικητικό ε, Συμβούλιο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ένα νούμερο ταυτοποίησης μέσω της νομοθεσίας μας εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι μια βάση για να προχωρήσουμε ή θα, θα έπρεπε να, αλλάξουμε βάση. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί έχουμε φτάσει σε μια καλύτερη χρονική στιγμή. Υπάρχουν περισσότερες προϋποθέσεις. Ε, μην ξεχνάμε και το LuxLeaks. Ε, χάρη στους δημοσιογράφους ε, έχουμε κάποια στοιχεία για να φτιάξουμε ένα ισχυρό εργαλείο. Δεύτερη σειρά ερωτήσεων. Έχουμε το Λουξεμβούργο και την Ελβετία. Υπήρξε μια αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο χωρών. Και πώς η, μια... η δράση του Λουξεμβούργου επηρεάζει την Ελβετία. Εμεί ασχολούμαστε πάρα πολύ με το Λουξεμβούργο και ξεχνάμε λιγάκι την Ελβετία σε όλη αυτή την ιστορία. Να ακούσουμε και μερικού ακόμα. Α, ξεχνάμε και μερικέ άλλε χώρε. Από το ECR, ο Μπέρντ Λούκε, αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω γερμανικά. Δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη αναφέρεται σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ζούντμαν. Πολύ ενδιαφέρον βεβαίως ε, η ιδέα των ενοποιημένων κερδών και η κατανομή τους στα κράτη αλλά Βεβαίω μιλήσετε για μια κλίδα κατανομής η οποία θα είναι οι πωλήσει. Κοιτάξτε, όπως το βλέπω εγώ, οι φόροι πρέπει να κατανεμηθούν ανάλογα με το κατά πόσο χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις που παράγουν υποδομές και άλλα τέτοια πράγματα. Γιατί οι φόροι είναι ακριβώς η τιμή για τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος ασφάλεια δικαίου, υποδομές, ε, δημόσια τάξη κτλ. Όλα αυτά, υγεία. Το να το κάνουμε ανάλογα με τις πωλήσει ε, θα οδηγήσει σε παράξενες ε, καταστάσεις. Ας πάρουμε π.χ. μια εξαγωγική επιχείρηση. Παράγει αγαθά και τα εξάγει όλα στο εξωτερικό. Και εμφανίζεται ως ένας διανομέας ας πούμε. Η πρότασή σας μετά δεν σημαίνει πως ε, οι φόροι θα πληρώνονται μόνο στο εξωτερικό. Παρά το ότι δεν χρησιμοποιούνται δημόσιες υπηρεσίες των ξένων χωρών για την παραγωγή. Το επόμενο ερώτημα αφορά το ζήτημα της δικαιοσύνης που ανέφερε ο κ. Μπελάμ και ήθελε να απαντήσει. Βεβαίως η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετρηθεί ακριβώς, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε είναι μια ισότητα της ε, φορολογίας ε, όταν έχουμε την ίδια φορολογητέα βάση. Και αυτό είναι μετρήσιμο. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πρέπει πραγματικά να περιμένουμε να υπάρχουν ε, κάποιοι ε, πληροφοριοδότες ή πως θα έπρεπε να έχουμε κάποιες υποχρεώσεις δημοσιότητας για τις ε, επιχειρήσεις έτσι ώστε από τα δημόσια δεδομένα να μπορούμε να διαβάσουμε ποια είναι τα κέρδη και ποιοι είναι οι φόροι που πληρώθηκαν. Μόνο αυτή την πληροφορία θέλουμε. Τα κέρδη και ποιοι ήταν οι φόροι που πλήρωσε συνολικά μια επιχείρηση. Αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν δυσκολίες ε, για να πούν ποια είναι τα κέρδη, αλλά θα έπρεπε νομίζω επί της αρχής να είναι δυνατόν να υπάρχουν κάποιες διατάξεις ε, του κράτους έτσι ώστε να υπάρχει μια ενιαία φορολογία, τουλάχιστον στο πλαίσιο ενός ε, ομίλου και να δούμε, όπως είπα, και ποιοι είναι οι φόροι που έχουν καταβληθεί. Σας ευχαριστώ, κύριος Τόρβαλτς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό το οποίο στη Φιλανδία λέμε το φαινόμενο της σαλαμοποίησης. Ε, το φαινόμενο του λουκάνικου, με συγχωρείτε, ότι όταν κάτι το ζουλάμε στο κέντρο, πρίζονται τα άκρα. Αν δηλαδή υποθέσουμε πως ε, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν ε, να καταλήξουν σε μια συμφωνία για να περιορίσουν τα παραθυράκια μέσω παραδείγματο χάρη της ε, κοινή φορολογικής βάσης τι θα συνέβαινε γιατί έχουμε ένα ασκιώδε ε, τραπεζικό σύστημα πιέζουμε λοιπόν στο κέντρο οπότε τι συμβαίνει τι θα συμβεί στα άκρα γιατί όπως είπε και ο καθηγητής ο κ. Ντόρφερ δεν ξέρουμε την έκταση τους, τους ε, τραπεζικού συστήματος νομίζαμε ότι το ξέραμε το 2007 αλλά είμαστε ακόμα σε χαρτογράφητα νερά και θα ήθελα να μου πείτε εσείς να κάνετε μία εικασία για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αν αλλάξουμε τους κανόνες. Ευχαριστώ. Ο Καθηγήτή Μπερλάν θα πρέπει να φύγει σε λίγα λεφτά, γι' αυτό να δώσουμε πρώτο το λόγο για να απαντήσει στις ερωτήσεις που αναφορούν και εν συνεχεία θα συνεχίσουν οι βουλευτέ με, με επιπλέον ερωτήσει. Θα είμαι πολύ σύντομο, Πρόεδρε. Γιατί θα αφήσω τους ε, συναδέλφους μου να απαντήσουν για τα στατιστικά στοιχεία, για τις λύσεις που ε, έχουν να προτείνουν. Δεν θέλω να σπετεριστώ τα χωράφια τους. Πρώτη παρατήρηση. Υπάρχει το άμεσο, το απτό πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή τώρα αμέσως για να καταπολεμήσουμε κάποιες πρακτικές που είναι όμως ε, το σύμπτωμα μιας αρρώστιας συστημικής, διαφορετικής. Ακούστηκε αυτό επίθετο. Και μπορεί να λυθεί με λύσεις Τη ενοποιημένη φορολογική βάση ή εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών. Γιατί το πρόβλημα από εκεί προέρχεται. Πολύ σωστά το είπατε στην αρχή, ότι συνεπάρχουν 28 διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα ε, και οι εταιρείε κυκλοφορούν ελεύθερα. Τώρα, ποια είναι η νομική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, η επίκαιρη νομική απάντηση. Υπάρχουν καταρχάς δυσκολίες λόγω της ύπαρξης ενός κράτους που ε, δίνει ruling, ε, πολιτικές συμφωνίες και δρά δηλαδή α, παράνομα και τι μπορούν να κάνουν τα άλλα κράτη απέναντι σε αυτό το πρώτο κράτος. Λοιπόν, αυτό που υπάρχει είναι αυτό που προτάθηκε το 1998 απέναντι στις τότε φορολογικές πρακτικές, της επιζημίες είναι ο, αυτό που είπε το Κομισιόν, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων. Δεν είναι η πανάκια, αλλά έχει λόγο ύπαρξης. Και γίνονται διάφοροι πειραματισμοί με τις κρατικές ενισχύσεις. Έχω κάποια όρια βέβαια στο τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το όπλο. Ε, το γαλλικό παράδειγμα για, τα, για το γοησκρή ας πούμε δεν μας πάει πολύ μακριά. Υπάρχει όμως δυνατότητα να καταπολεμήσουμε, και αυτό έγινε και στο παρελθόν, κάποιες πρακτικές ή καθεστώτα, γιατί άλλο πρακτικές έχουν καθεστώτα, και πιο συχνά τα καθεστώτα που δημιουργούν τα κράτη παρά οι διοικητικέ πρακτικές που μπορούν να καλυφθούν με τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Και αν θέλουμε να φτάσουμε σε πιο καινοτόμε απαντήσεις είναι τι μπορούν να κάνουν τα άλλα κράτη απέναντι σε κρατικέ που θεωρούν επιζήμιες. Είχαμε την αντίδραση του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών όπου είπε οι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε στο Λουξεμβούργο να κάνουν ό,τι γουστάρουν, εγώ θα τις φορολογήσω στη Γαλλία και έτσι θα καλύψω, θα εισπράξω τη διαφορά. Εντάξει, ηθικός πώς το καταλαβαίνω, αλλά νομικός πώς η απάντηση ε, είναι μετρημένη, γιατί το δίκαιο της Ένωσης θέτει όρια σε τέτοιες αντιδράσεις προς το παρόν. Προς το παρόν. Και η νομολογία του δικαστηρίου δείχνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε απέναντι σε κράτη τα οποία έχουν μια φορολογία πιο πλεονεκτική, πιο ευνοϊκή. Και η Ιρλανδία το είχε καταλάβει στο παρελθόν. Την επικρίναμε, ας πούμε, για τα docs του Δουβλίνου, ας πούμε, και είχε ένα καθεστώς για όλες τις εταιρείε 12%. Και τελικά δεν λέμε τίποτα πια επ' αυτού, ε. Τι άλλο να πούμε. Υπάρχουν απαντήσεις που μπορούν να δοθούν, αλλά που θα πρέπει να ελεγχθούν σε ό,τι αφορά την νομιμότητά τους απέναντι στο δίκαιο της Ένωσης. Κατά τα λοιπά, δύο προτάσεις πριν σας εγκαταλείψω, δυστυχώς. Η μία από τις λύσεις είναι, αφορά το μέλλον και όχι το παρόν. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που υπόθηκαν για την ενωπημένη βάση του φόρου των επιχειρήσεων. Αυτό που θα μπορούσε να εξετάσουμε, δεν ξέρω σε ποιο πλαίσιο βέβαια, πέρα από την οδηγία για τη διαφάνεια, για τα ρούλη, η οποία είναι απαραίτητη φυσικά, είναι να εισάγουμε σε μια οδηγία αυτό που εισάγαμε στην οδηγία για την φορολογία των καταθέσεων, δηλαδή την, πραγματική, την αρχή της πραγματικής φορολόγησης μπορεί κανείς να πάει δεξιά και αριστερά και να ε, επωφεληθεί από πιο ευνοϊκούς ε, φορολογικούς συντελεστές ε, υπό τον όρο ότι υπάρχει πραγματική φορολογία σε κάποιο κράτος τελικά. Ποιο κράτος τώρα, ποιο κράτος. Αυτό είναι το θέμα της ιδέας που ακούστηκε για την κατανομή της φορολογίας. Υπάρχουν ε, κλίδες κατανομής που υπάρχουν στην οδηγία για τους φόρους, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Υπάρχει βέβαια και το πρόβλημα των εργαζομένων. Εδώ λαμβάνουμε υπόψη μας ποια είναι η δομή στα κράτη-μέλη για να κατανείμουμε τη φορολογητέα βάση. Και μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη λύση με την ιδέα που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Να επαθαληθεύσουμε δηλαδή ε, αν τα κράτη το παρακάνουν ε, στην προσπάθεια να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Γιατί θέλουμε τελικά να προσπαθήσουμε για μια συγκεκριμένη εταιρεία, ας πούμε, Χ, να υπάρχει μια ισορροπημένη κατανομή της φορολογίας, έτσι. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με, με ομίλους. Αυτά δεν τα λέω τώρα σε δεοντολογικό επίπεδο, σε επίπεδο ηθικής, αλλά σε επίπεδο νομικό. Είμαι έτοιμος φυσικά να απαντήσω και γραπτός σε όλες τις ερωτήσεις, σε όλα τα, τα θέματα που τέθηκαν. Ε, πρέπει αναγκαστικά να σας εγκαταλείψω για λόγους ανεξάρτητους θέλησής μου και σας ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, καθηγητά. Και θα παραμένουμε... και θα παραμείνουμε σε επαφή. Λοιπόν. Έχω ε, να συνεχιστεί ο κατάλογος των ομιλητών και οι δύο πλέον εμπειρογνώμονες θα απαντήσουν σε όλα. Καταρχήν για την Γουέ Ματίας. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πολλές ερωτήσεις που έγιναν ήδη από άλλους συναδέλφους. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, μιλήσαμε ήδη για την προσέγγιση της ε, φοροαποφυγής, αλλά τώρα μπαίνουμε σε άλλα χωράφια με όλα αυτά τα προβλήματα που δημοσιοποιήθηκαν περνάμε σε μια νέα προσέγγιση που σχετίζεται με το ότι Φαίνεται πως η φοροαποφυγή βασίζεται στην διαφάνεια. Αυτή είναι νομίζω η νέα βασική προσέγγιση και λαμβάνουμε υπόψη εδώ πέρα πως η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών θα μειώσει την φοροαποφυγή σε φορολογικούς παραδείσους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε πως αυτή είναι η καλύτερη προσέγγιση. Και αν όχι, ποιοι είναι οι περιορισμοί που έχει και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Ξέρω πως ο κύριος ε, Σίγμουντ το ανέφερε αυτό το ζήτημα στην δημοσίευσή του του 2004 με τον κύριο Γιωχάνσεν για τις συστάσεις των G20. Μιλάτε παραδείγματο χάρη για για κάποιον φόρο είτε στις διάφορες προσόδους, είτε στην ε, πηγή και με κάτι άλλο πάρα πολύ συγκεκριμένο, γιατί η Ελίζα μίλησε για διάφορες ε, δικαιοδοσίες και το ανέφεραν κι άλλοι. Ως ερευνητές εσείς όταν κάνετε την έρευνά σας, που θεωρείτε ότι λαμβάνουν χώρα οι οικονομικές δραστηριότητες, ε, στην ε, υπεράκτια τοποθεσία ή σε άλλες δικαιοδοσίε. Είναι σημαντικό νομίζω και αυτό να το ξέρουμε. Το πρόβλημα Nexus. Ευχαριστούμε Μαρίσα. Pour le FDD, Ο Μάρκο Βάλλη από το FDD. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τους τρεις ομιλητές και τον ομιλητή που μόλις μας έφυγε. Βασικά για αυτόν είναι η, ερώτηση. Με τον κύριο Κίντορφ ε, συμφωνώ το βασικό πρόβλημα είναι η διαφάνεια. Αλλά είμαι απογοητευμένος από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το σκάνδαλο. Βλέπουμε το σκάνδαλο, αποκαλύπτεται με τα LuxLeaks, κινητοποιούνται όλοι ...κοινοποιούνται γιατί αγανακτούν όλοι οι πολίτες, οι οποίοι πλήττονται από αυτήν την κατάσταση, η οποία είναι παράδοξη. Γίνεται μια οδηγία, η οποία θα έπρεπε να μας εξασφαλίσει την διαφάνεια, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η οδηγία είναι απλούστατα ένα φύλλο οικής για να βουλώσουμε τα στόματα όλων αυτών που προσπαθούν να εξασφαλίσουν λίγη ηθική, δεοντολογία, διαφάνεια κτλ. Απλώς για να βουλώσουμε τα στόματα. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της οδηγίας, τουλάχιστον ε, μιλάμε για το πρόβλημα έλλειψης διαφάνειας μεταξύ των κρατών, γιατί κρατάνε τα μυστικά τους. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στο Κοινοβούλιο για να τροποποιήσουμε αυτή την οδηγία. Εμείς και η Κομισιόν δηλαδή, εν πάση Κάτι την άποψή Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Υπάρχουν άλλοι προβουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο στα πλαίσια του Catch Ο κύριος Κίρτσος. Ευχαριστώ. Μιλάμε για το Λουξεμβούργο και την Ελβετία, αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη των ειδικών για τις πέντε άλλες χώρες μέλη που έχουν το πιο επιθετικό φορολογικό καθεστώς όσον αφορά την φοροαποφυγή. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Έχουμε τον κύριο Σάιμον. Απέναντί μου είστε. νότ. Ανιστότς. Αυτοί οι δύο μόνο. Ο Πίτερ. Μια ερώτηση προς τον κύριο Ντέρφερ. Δεν χρειάζεται νομίζω να βάλει τα ακουστικά. Αν σας ψάξει κανείς στο Google ε, βλέπει τις δημοσιεύσεις σας. Στη δουλειά σας λοιπόν, τι είχατε, ε, είδατε ποτέ αυτό το οποίο ήρθαν και μας είπαν εδώ πέρα διάφοροι εφοριακοί. Ότι δηλαδή ένα πρόβλημα εντός των φορολογικών διοικήσεων είναι η έλλειψη προσωπικού αλλά και εντός των αρχών υπάρχουν κάποια όρια πάνω στα οποία προσκρούν οι εφοριακοί. Δηλαδή λένε πως ε, μία μονάδα ε, κάνει τις φορολογικές συμφωνίες και οι απλοί ας πούμε εφοριακοί δεν μπορούν πια να μπουν σε αυτήν την επιχείρηση. ισχύει αυτό, δηλαδή ότι υπάρχουν ξεχωριστές μονάδες των φορολογικών διοικήσεων που κάνουν αυτές τις ε, συμφωνίες. Εσείς ε, είδατε τέτοια πράγματα, υπέψαν τέτοια πράγματα στην αντίληψή σας. Σας ευχαριστώ, Ανελίζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές και τον τρίτο ομιλητή που έφυγε. Μας βοήθησατε με τα σχόλιά σας. Έχω μία ερώτηση για την ενοποιημένη φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Φυσικά, για μας τους σοσιαλιστές είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όμως υπήρχαν πάρα πολλά εμπόδια για να υιοθετηθεί, όπως αναφέρθηκε ήδη. Διερωτώ με, μπορείτε να σχολιάσετε γιατί συνέβη αυτό. Φυσικά το μοντέλο της ενωπημένης βάσης που είχε προτείνει το Κοινοβούλιο ήταν αρκετά περίπλοκο. Δεν αφορούσε μόνο τις ε, πωλήσει, αλλά είχε και άλλα στοιχεία στην εξίσωση. Αντίθετα από αυτό που αναφέρθηκε πριν. Γιατί υπήρξαν αυτά τα εμπόδια για να υιοθετηθεί η πρόταση αυτή και γιατί δεν ήταν ε, βασικό στοιχείο του προγράμματος του ΩΣΑ ε, κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς των κερδών, δεδομένου ότι η προσέγγιση στη φορολογική βάση που έχουμε σε αυτό το CCTV, δηλαδή την ενωπημένη φορολογική βάση, έχει γίνει αποδεκτή ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα επίσης, αν μου επιτρέπετε, ε, μετά την συνεδρίαση και αφού σκεφτούμε αυτά που μας πείτε, να μας δώσετε την ευκαιρία να, σας, να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και να σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα. Τώρα, ο Πρόεδρος θα κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις και θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας. Καταρχάς, ακούστε. Να απαντήσω σε κάτι που είπε ο καθηγητής Μπέρλα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε κάποια προσφυγή ενό κράτου μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή του, ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καμία προσφυγή. Σίγουρα νομικός πώς Στις περισσότερες περιπτώσεις κανένας νόμος δεν παραβιάζεται και κυρίως κανένας κοινοτικός νόμος. Εκτός από την, τις κρατικές ανισχύσεις και το δίκαιο φορολογικό ανταγωνισμό. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν ξεκινήσει ε, έναν αγώνα να, για να κλέβουν τη φορολογική βάση του γειτονά τους. Και αυτό είναι κατά της φορολογικής δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά, κανένα δεν θέλησε να κάνει νομολογία το δικαστήριο και το γεγονός αυτό πραγματικά με εκπλήσει. Όταν απευθυνόμαστε στις υπηρεσίες μας, τις νομικές, είναι εδώ οι πρόσωποι της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, που είναι και η καλύτερη νομική υπηρεσία όλων, πάντα μας λέει έτσι πολύ προσεκτικά και συνετά, α, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Μου κάνει εντύπωση, εν πάση αυτό. Μία παρατήρηση για την αρχή της πραγματική και αποτελεσματικής φορολόγηση. Την περασμένη εβδομάδα ήρθαν εδώ αυθόρμητα, και το εκτιμήσαμε, ο, οι πρωθυπουργοί του Ζέρση και Γκέρνσι και πρότειναν να συμμετάσχουν στην έρευνα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Και αμέσω του απευθύναμε το ερωτηματολόγιο που στείλαμε και στα υπόλοιπα 28 κρατημένα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εκπρόσωπο λοιπόν του Τζέρσι και του Γκέρνσι στις Βρυξέλλες μας είπε με θαυμάσιο τρόπο ότι είμαστε υπέρ τη αρχή της πραγματικής φορολόγηση που ανέφερε και ο καθηγητής Μπέρλα. Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη έδρα σε μας, θα διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που φτάνουν σε μας ε, έρχονται αφού πρώτα καταβληθεί ο φόρος που έπρεπε να καταβληθεί στη χώρα που έπρεπε. Και πληρώνεται και ο φόρος για, με, αφού ελέγξουμε που έχουν γίνει οι πραγματικές επενδύσεις. Οπότε είμαστε άμεμπτοι. Και πρέπει να ξέρετε βέβαια ότι σε εμάς δεν υπάρχει καμία φορολογία. Αυτό το λέω ανεκδοτολογικά. Το, και το λέω έτσι με διάθεση σκοπτική. Το ερώτημα είναι, ποιο επαληθεύει ότι υπάρχει πραγματική φορολόγηση στο πολιτικονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη παρατήρηση. Το είπα προηγουμένως. Είναι μια ερώτηση της Μαρίζας που με αναγκάζει να την το ψάξω περισσότερο. Είναι το θέμα του apportionment. Το θέμα της κατανομής. Της, ε, εδώ έχει να κάνει με την ε, ψηφιακή οικονομία. Ε, πριν από δύο χρόνια στο, στη Γερουσία των ΗΠΑ έγινε, έγινε μία ακρόαση για την εταιρεία Apple. Apple δηλαδή. Ο γερουσιαστής Καρλ Λέβιν, πρόεδρος της, υποεπιτροπής, της Εξεταστικής Επιτροπής υπεύθυνη να ερευνήσει τις φορολογικές πρακτικές των Αμερικανικών πολυεθνικών, ο κύριος Κουκ, ο διευθυντής της Apple, είπε ότι η εταιρεία του πλέει στα σύννεφα τις νεφέλες. Δημιουργεί αξία, αλλά δεν είναι εύκολο, είναι αδύνατο μάλλον να εντοπίσει την αξία που δημιουργείται, την υπεραξία που δημιουργείται. Και άρα τι να φορολογήσεις. Ε, εν πάση περιπτώσει, ε, το cloud, το, το, το νέφος της Apple αγνοεί βεβαίως τις τέσσερις υπόλοιπες υπήρους και ασχολείται μόνο με την Αμερικανική, αλλά και εκεί ακόμα δεν μπορεί να εντοπιστεί. Να σας πω κάτι άλλο τώρα. Ο έχει θεσπίσει κανόνες που παρακολουθούν και δέχονται πολλές ε, φορολογικές αρχές μας. Και πρότεινε μάλιστα στον ΠΕΠΣ του να τις επικαιροποιήσει. Οι χώρες όμως που συμμετέχουν έχουν μια σημαντική εμπειρία για αυτό το πρόβλημα ε, κατανομής της φορολογικής βάσης. Οι Ηνωμένε Πολιτείε επίσης έχουν ένα ομοσπονδιακό φόρο για τις εταιρείες του και 100 χρόνια πάνω από 40 πολιτείες προσθέτουν και πολιτιακό φόρο. Μία εταιρεία λοιπόν, η οποία έχει δραστηριότητα σε περισσότερες από μία πολιτείες, έχει αυτό το πρόβλημα σε ποια πολιτεία τελικά θα πρέπει να φορολογηθεί. Ή εν πάση πώ ε, κατανέμεται η εν παση πως κατανεμεται η φορολογικη της βάση μεταξύ των πολιτιών. Μια και κάθε πολιτεία έχει διαφορετικό φορολογικό σύστημα. Είτε το apportionment, είτε άλλο σύστημα. Υπάρχει νομολογία του Αντάτου Δικαστηρίου του Αμερικάνικου. Μπορεί να μας χρησιμεύσει ως βάση. Στον Καναδά είναι το ίδιο. Σε μια χώρα ομοσπονδιακή όπως η Ελβετία υπάρχει επίσης ε, η φορολογία των καντονίων. Και ίσως από εκεί θα μπορούσαμε να ενταχτούμε κάποια πράγματα. Ποια είναι η εντύπωση που έχετε λοιπόν για όλες αυτές τις, α, για αυτά τα φορολογικά καθεστώτα. Uh, Θα ήθελα να ξεκινήσω με το παράδειγμα αυτό του Λουκάνικου γιατί πραγματικά ήταν πολύ εύγλωτο. Ναι, ναι, είναι στο μυαλό του κάθε Γερμανού. Κοιτάξτε, εγώ είμαι και Εβραίος, δεν μπορεί να έχει χειρινό μέσα το Λουκάνικο, εν πάση Το παράδειγμα σε ισχύει μόνο για Λουκάνικα μαλακά, όχι σαλάμια. Άμα γίνει πιο σκληρό λοιπόν, δεν λειτουργεί έτσι όπως είπατε. Και έτσι απαντάμε στο δικό σας το ερώτημα. Σε τι ωφελεί αυτή η διαφάνεια. Δεν θεωρώ πως λύνει το πρόβλημα αυτό καθεαυτό. Αλλά καθιστά την φοροδιαφυγή πιο ακριβή. Έχουμε π.χ. το καθεστώς ε, ανταλλαγής ε, δεδομένων, ήδη έχει υπογραφεί από κάποιους, θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες το 16 και 17. Ο Παναμάς δεν θα το υπογράψει, αλλά θα διαλέξει κάποια πράγματα και θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να αυξήσει τις τιμές ε, και τα τέλη για να έχει κανείς λογαριασμό στον Παναμά. Και βεβαίως ε, ένα άλλο θέμα είναι η ανταλλαγή ε, δεδομένων για τους υπηκόους. Δηλαδή, αν μια γερμανική τράπεζα ζητήσει από μια συγκαπουριανή τράπεζα τα δεδομένα ενός γερμανού υπηκόου, είναι εύκολο να παρακαμφθεί αυτό μέσω ενός ε, άλλου ενδιάμεσου ο οποίος θα έχει άλλη Αλλά και αυτό κοστίζει. Και υπάρχουν άλλα μέτρα για να παρακαμφθεί αυτό. Να αγοράσει κανείς ε, χρυσό, ακριβά αυτοκίνητα, τέχνη. Και ε, πού μπορεί κανείς να αποθηκεύσει τέχνη. Στο Λουξεμβούργο, παραδείγματος χάρη, φτιαχτεί ένα καινούριο τέρμιναρ για αυτή τη δουλειά. Είναι ανώνυμο λοιπόν, αλλά κοστίζει, είναι επικίνδυνο, οπότε το λουκάνικο αρχίζει και σκληραίνει. Και γίνεται δυσκολότερο να αποφύγει κανείς τον φόρο. Οπότε κάποια πρόοδος είναι και αυτή και νομίζω πως μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Ε, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα ε, άπαξ και διαπαντός, αυτό είναι αδύνατον αλλά μπορούμε να έχουμε κάποιες σταδιακές βελτιώσεις. Κάτι άλλο, ναι κύριε Πρόεδρε, το αναφέρατε. Και εμένα μου προξένει η εντύπωση ότι χρειάστηκε η Κομισιόν τόσο χρόνο για να σκεφτεί το να χαρακτηρίσει αυτές τις αποφάσεις ως παράνομες επιδοτήσεις γιατί είναι απολύτως λογικό και έπρεπε να έχει γίνει πριν από 20 χρόνια αλλά ε, χρειάστηκαν 20 χρόνια και δεν νομίζω πως έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση ο κύριος Τόιρερ ρώτησε για την βιομηχανία αυτή της φοροαποφυγής, τον κλάδο αν θέλετε είναι ένας καλός ορισμός και χαρακτηρισμός γιατί υπάρχει μία παράλληλη κοινωνία η οποία αναπτύσσεται όχι κοινωνία με την πολιτισμική έννοια αλλά με την έννοια πως έχουν τους δικούς τους νόμους για τη φορολογία είναι μία αυτοσχέδια φορολογία της ε, κλίμακας φορολογία εισοδήματο και βεβαίω καταστρέφει οποιαδήποτε πολιτισμένη κοινωνία. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό ο παράλληλο μηχανισμό. Κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι άλλο ένα επιχείρημα για να γίνουν απλούστεροι οι φορολογικοί κώδικες για να μην είναι μόνο ειδικοί αυτοί οι οποίοι τα καταλαβαίνουν και μπορούν να πουλήσουν αυτή τη γνώση μετά σε όποιον πληρώνει τα περισσότερα. ή μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε ολόκληρο το σύστημα. Την σχέση δηλαδή μεταξύ των διαφόρων ειδών φόρων. Ίσως θα ήταν καλύτερο να έχουμε ψηλότερο ΦΠΑ γιατί είναι ένας φόρος στην πηγή και ταυτόχρονα να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος για να και να μην αποφεύγεται, να γίνει πιο δύσκολη η αποφυγή του. Ίσως αυτό χρειάζεται, δηλαδή να έχουμε υψηλότερο φόρο εκεί όπου είναι εύκολο να ε, συλλεγούν και λιγότερο εκεί όπου είναι πιο δύσκολο. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ. Ah, your question. <laughs> Uh, για να δω... Ε, επιγραμματικά, επιγραμματικά. Μίλησα για αυτό το οποίο μας είπαν οι φορολόγοι, εφοριακοί και κάτι άλλο εκτός μικροφώνου. Ναι, ναι, σωστά, οι εφοριακοί Αυτό το ακούω συχνά από τα συνδικάτα των εφοριακών ότι χρειάζονται προσωπικό. Και πάντα αναρωτιέμαι χρειάζονται περισσότερο προσωπικό για να κυνηγήσουν αυτούς που αποφεύγουν τους πολλούς φόρους αφού τελειώσουν με αυτούς που βγάζουν λίγα. Αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι περισσότερη εφοριακή αλλά καλύτερη, πιο καταρτισμένη. Στο κρατήδιο της ΕΣΥΣ προς τα εκεί πάνε. Πριν από δύο χρόνια υπήρξε μια ανακοίνωση τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών του Κρατηδίου της ΕΣΥΣ και έλεγαν πως έχουν τώρα κάποιους ειδικευμένου νομικούς και τους ρώτησα πόσοι είναι, αν δουλεύουν με πλήρες ωράριο και αν έχουν κάποια επιτυχία. Δεν μου απάντησαν. Ξαναρώτησα δύο χρόνια μετά, πάλι καμία απάντηση. Οπότε τίποτα δεν έχει γίνει. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ταυτόχρονα με τους 8 αυτούς ανθρώπους στην ΕΣΥ. Οι τέσσερις μεγάλες λογιστικές εταιρείε έχουν 9.000 υπαλλήλους στο κρατήδιο της ΕΣΥ πάντα. Οπότε δεν χρειάζεται πάλι να αρχίσουμε να κυνηγάμε όποιον πουλάει τυρόπιτες ή λοκάνικα στην ΕΣΥ χρειαζόμαστε καταρτισμένους ανθρώπους, εκατοντάδες, για να μείνουν τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τις ε, τέσσερις μεγάλες λογιστικές εταιρείες. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much for, for all the... Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Ακούστηκαν πολλές ερωτήσεις για το CCTB, την ενοποιημένη φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Καταρχάς δεν υπάρχει τέλειος μαθηματικός τύπος για να φορολογήσουμε τα κέρδη. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να φορολογήσεις τα κέρδη των πολυεθνικών. Με τις μεταβιβαστικές τιμολογήσεις και αυτό που κάνουμε στην, όπως κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το apportionment. Ξεκινάς δηλαδή από τα ενοποιημένα κέρδη και μετά με ένα τύπο ε, κάνεις μια κατανομή της φορολόγησης. όλες, όλα τα ομοσπονδιακά κράτη δεν χρησιμοποιούν ε, το transfer pricing, χρησιμοποιούν το apportionment. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει και να κινηθεί. Πώς μπορείς να φορολογήσεις τα κέρδη, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν τη δική τους μορφή apportionment που σύν χρόνο οδήγησε σε έναν τύπο που βασίζεται περισσότερο στις πωλήσει. Δηλαδή έτσι φορολογούν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, Καλιφόρνια, Νιου Τζέρσι, όλες ε, οι πολιτείες, περισσότερες χρησιμοποιούν ένα, μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο apportionment που, που βασίζεται στις πολιτείες και τους βολεύει, είναι ικανοποιημένοι. Φυσικά πρέπει να διδαχτούμε γιατί είναι ικανοποιημένοι με αυτό το σύστημα. Είναι ικανοποιημένοι γιατί αν χρησιμοποιήσουμε τις πολιτείες τότε ε, βλέπεις πού γίνονται οι πωλήσει. Ε, και δεν υπάρχει περίπτωση οι εταιρείε να πούνε ψεύτικο τόπο όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ε, γιατί μπορεί να στείλει εύκολα τα κέρδη σου στη Βερμούδα, αλλά δεν μπορεί να στείλει του πελάτε σου στη Βερμούδα, έτσι. Οι πελάτε είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Νιου Τζέρζι, η Καλιφόρνια και δεν μπορεί να του μετακινήσει. Μπορεί να σκεφτεί πιο περίπλοκου τύπου αυτό που υπάρχει στο σημερινό σχέδιο για το CCTB, όπου το κέρδη σου, ε, ε, μάλλον φορολογείς όχι μόνο με βάση τις πωλήσει, αλλά ε, και το που βρίσκεται το φυσικό σου κεφάλαιο λοιπά. Κάνα πρόβλημα. Έτσι όμως αφήνεις κίνητρα ε, στις εταιρείες να μετακινήσουν τα εργοστάσια τους, τις πραγματικές δραστηριότητες τους σε χώρες όπου οι φόροι είναι χαμηλοί. Ενώ αν έχουμε ένα σύστημα που να, βασίζεται στις πολίτες, δεν γίνεται ε, κάτι τέτοιο. Ας πούμε, η Ιρλανδία μπορεί να κρατήσει το 12% εταιρικού φόρου, αλλά δεν έχει κανένα κίνητρο, ας πούμε, οι εταιρείε να έχουν εταιρική έδρα ή το εργατικό του δυναμικό στην Ιρλανδία. Γιατί τα κέρδη θα είναι ένα τμήμα μόνο ε, του κομματιού που γίνονται οι πραγματικές πωλήσει, έτσι. Και αυτή είναι η ομορφιά αυτού του συστήματος. Ποιο είναι το, πρόβλημα με τη μετακίνηση της πραγματικής δραστηριότητας α, της επιχείρησης εκεί που έχουμε χαμηλούς φόρους. Τι νόημα έχει αυτό. Ποιο είναι το καλό Τι καλό κάνει ο φορολογικός ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 12,5% του, της Ιρλανδίας, ας πούμε, τι καλό κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να προστατεύουν ε, τις επιχειρήσεις από να τις εκμεταλλεύονται κάποιες κυβερνήσεις, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα, κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να λέει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει στοιχείο που να, που δικαιολογεί αυτή την θέση. Ακούστηκαν πολλές ερωτήσεις για τη διαφάνεια. Καλή η διαφάνεια. Τι σημαίνει όμως. Ένας τρόπος για να έχεις διαφάνεια είναι να γίνεται κάποια ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτόματη, ας πούμε, ανταλλαγή πληροφοριών πληροφοριών για τα τραπεζικά δεδομένα. Πού θα γίνει η πραγματικότητα μεταξύ των ε, μεγάλων οικονομιών μέχρι το 2018 ή αυτόματη ανταλλαγή των φορολογικών συμφωνιών. Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά μερικές φορές αυτό δεν ε, λύνει το βασικό πρόβλημα της διαφάνειας που είναι το μπορούμε να ξέρουμε ποιος κερδίζει τι και το αν ο κόσμος πληρώνει φόρους με βάση την, την ικανότητά του να τους πληρώσει, το δυναμικό του, το, την περιουσία του. Η ενσωμάτωση της έννοιας της η θα ήταν ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό μητρό ή οικονομικό μητρό. Και εκεί όλα τα ομόλογα, όλα τα πάτα παράγωγα, ε, όλοι οι τίτλοι, κινητές αξίες κτλ. Ε, καταγράφονται όπως κάνουν, ας πούμε, κάνουμε στο κτηματολόγιο επί αιώνες. Αυτά τα μητρώα δημιουργήθηκαν πριν από αιώνες σε πολλές περιπτώσεις, όπου ο βασικός πλούτος, ας πούμε, έγκυας περιουσίας, δημιουργήθηκαν μάλιστα από τα τέλη του 18ου αιώνα και όπου καταγράφονται όλοι οι πλούσιοι ή ο πλούσιος του καθενός. Ε, σήμερα ε, ο πλούτος των περισσότερων δεν είναι η έγκυα περιουσία, αλλά είναι ο χρηματοπιστωτικός πλούτος. Τέτοιου τύπου μητρώα χρηματοπιστωτικά υπάρχουν, αλλά τα ε, διαχειρίζονται τα κεντρικά αποθετήρια, δηλαδή, που είναι ιδιωτικά, έτσι. Ούτε οι αφορίε ε, τα διαχειρίζονται, ούτε οι στατιστικέ υπηρεσίε δεν χρησιμοποιούνται για στατιστικέ υπηρεσίε, ούτε παρακολουθούμε την, ε, τη σταθερότητα. Θα μπορούσαν αυτά τα μητρώα που υπάρχουν, τα κεντρικά αποθετήρια αυτά που υπάρχουν, να χρησιμοποιηθούν για όλα αυτά τα πράγματα. Επομένω, ε, καλή είναι η διαφάνεια, αλλά τι εννοούμε με αυτήν. Ανταλλαγή των πληροφοριών, αυτή δεν είναι αρκετή. Και θα υπήρχε τέτοια διαφάνεια αν είχαμε ένα τέτοιο παγκόσμιο μητρό που θα καταγραφόταν όλο ο χρηματοοικονομικός πλούτος. Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί τα κράτη που χάνουν ε, το φορολογικό τους πλούτο, τα φορολογικά τους έσοδα, γιατί δεν παραπονούνται, γιατί δεν κάνουν προσφυγή. Ε, Ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια αυτό το πράγμα και όμως υπάρχουν ελάχιστες προσφυγές από κράτη-μέλη που είναι θύματα τέτοιων πρακτικών. Ένας λόγος είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία. Γιατί δεν υπάρχει ακριβώς αυτό το αρχείο που σας περιέγραφα. Εάν δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η φορολογική απώλεια λόγω της φοροδιαφυγής ή φοροδιαφυγής, τότε πώς να παραπονεθείς, πού να προσφύγεις. Ένας άλλος λόγος είναι ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει επαρκώς ότι υπάρχει μια απλή λύση στο πρόβλημα αυτό. Πού είναι. Εάν κάποια κράτη θέλουν να κλέψουν ε, τα φορολογικά έσοδα των γειτόνων τους, τα θύματα, τα κράτη θύματα θα πρέπει να ε, επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις ανάλογα με την απώλεια που έχουν λόγω της κλοπής αυτής των φορολογικών εσόδων. Τι είδους κυρώσεις θα μπορούσαν να επιβάλλουν με ρεαλιστικό τρόπο. Είναι ε, φορολόγηση στην πηγή. Αν μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Λουξεμβούργο φερειπή, αρνηθεί να συνεργαστεί με κάποιες σημαντικές χώρες είναι απόλυτα δυνατόν τα άλλα κρατημέλη να πούνε «Α, κάνε αυτό που θέλεις, να τι μας κόστισε, τι διαφυγόντα έσοδα είχαμε, επομένως τα αντίπεινα ποια είναι, παρακρατούμε το φόρο σε διασυνοριακές ε, οικονομικές συναλλαγές. Άλλος τρόπος είναι οι δασμοί. Φυσικά αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αναλογικοί με το διαφυγόν κέρδος. Δηλαδή με τις πρακτικές αυτές που κάνει Φερρυπίν το Λουξεμβούργο. Να, γιατί χρειαζόμαστε λοιπόν στοιχεία για να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε το διαφυγόν φορολογικό έσοδο. Εν συνεχεία, αφού ξε... μάθουν όλα ποιο είναι αυτό το διαφυγόν έσοδο, τα διαφυγόντα έσοδα, έχει νόημα μια πια προσέγγιση. Μάλιστα. Όλα αυτά βέβαια δείχνουν και την τεράστια δυσκολία. Προηγουμένως σας μίλησα για την αρχή της καλής πίστης μεταξύ χωρών μελών. Βέβαια όλες αυτές οι μέθοδοι θα εφαρμόζονταν μόνο αν υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές ε, αντίληψης μεταξύ χωρών μελών. Πολύ δύσκολα όλα αυτά, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, να σας πω μόνο το εξής. Για το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Το περίεργο στην περίπτωση της Ιρλανδίας δεν είναι το 12,5%. Εξάλλου κανείς δεν ξέρει τον παρονομαστή του. Εφόσον δεν έχουμε συμφωνήσει για το CCCTB. Οι Ιρλανδοί τα υπολογίζουν όπως θέλουν αυτά. Έχω δει τις συγκρίσεις που κάναν μερικές επιχειρήσεις που λένε ότι το 12,5% στην Ιρλανδία καταλήγει σε υψηλότερο φόρο από ότι το 28 ή 30% σε άλλο κράτος μέλος όπου ορίζεται αλλιώς η φορολόγηση. Δεν είναι το 12% λοιπόν το πρόβλημα αλλά το 1%. Η κοινωνία Adobe με 500 εκατομμύρια ευρώ κέρδος τον περασμένο χρόνο πραγματοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πραγματοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε 3 εκατομμύρια σε φόρους. Αν είχε πληρώσει το 12,5% θα λέγαμε εντάξει ο ανταγωνισμός. Όχι, όλα αυτά βασίζονται σε ψεύδι και αυτό πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ τώρα. Σας προτείνω να ευχαριστήσουμε τους ομιλητάς. Θα μείνουμε σε επαφή μαζί τους, ιδιαίτερα οι συντονιστές. Έχει λήξει η μερίσια διάταξη και λέω να κλείσει και η συνεδρίαση, αλλά να μείνουν στην αίθουσα τα μέλη της αντιπροσωπείας που από αύριο θα εποπτεύσουν στο Βέλγιο για να... Α, ο Μιχαήλ θέλει κάτι να πει. Μετά, από όταν τελειώσω. Η Ελίζα πρέπει να φύγει τώρα και οι συντονιστές φυσικά παίζουν βασικό ρόλο για την αποστολή αυτή στο Βέλγιο. Ο Μιχαήλ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιες παρατηρήσεις ε, των συνεισηγητών. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, λέει ο πρόεδρος. Νομίζω πως αυτά τα οποία είδαμε σήμερα κατέστησαν σαφές το πόσο σημαντικό ήταν να καλέσουμε αφενός τους δημοσιογράφους είδαμε πως ε, δεν θα συζητούσαμε τόσο πολύ το θέμα της ε, φοροαποφυγής αν δεν υπήρχαν οι δημοσιογράφοι. Εγώ λοιπόν ως σημερινό, σημερινό συμπέρασμα βγάζω το ότι ε, υφίστανται τεράστια πίεση οι δημοσιογράφοι και αυτοί οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες και πρέπει να κάνουμε κάτι για να τους προστατεύσουμε καλύτερα γιατί το ακούσαμε αυτό από μια προσωπική τραγωδία δύο ανθρώπων απόψε το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση πρέπει λοιπόν να το έχουμε ψηλά νομίζω στις προτεραιότητες μας και νομίζω πως ο καθηγητής ε, Μπερλάν δεν είναι τόσο αισιόδοξο ότι μπορούμε να δούμε το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε με ένα νομικό πλαίσιο και οι κύριοι Ντέρφερ και Τσούγκμαν μίλησαν για την διαφάνεια η οποία δεν επαρκεί οπότε μας είπατε κάποια πράγματα για το τι μπορούμε να κάνουμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ειδικούς και είμαι σίγουρος πως θα πρέπει να ερευνήσουμε πιο πολύ τους μηχανισμούς των ενδομηλικών συναλλαγών και τις άλλες ε, προτάσεις που ακούσαμε να περάσουμε από τον εταιρικό φόρο στο ΦΠΑ είναι μια ιδέα κύριε Πρόεδρε που θεωρώ πως θα πρέπει να την συμπεριλάβουμε και να συμπεριλάβουμε και την πρόσκληση κάποιων ειδικών την φορολογία για να δούμε τα διάφορα μοντέλα ε, νέων συστημάτων φορολογίας ε, ε, που θα περιλαμβάνουν και την μετατόπιση σε μια παγκόσμια ψηφιακή οικονομία. Αυτά τα ολίγα από μένα και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους εμπειρογνωμονές μας. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπες. Ελίζα, ναι. Σύντομα σύντομα. Συμμερίζομαι και εγώ τα συμπεράσματα του Μιχαήλ. Επί τριών θεμάτων. Πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μίλησαν και θα ήθελα να συνεχιστούν οι επαφές. Δεύτερον, απόλυτη ανάγκη να ληφθούν πολιτικά μέτρα σε πανενωσιακό επίπεδο για να προστατευτούν οι πληροφοριοδότες. Με έμπνευση ίσως στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και ε, επίσης νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε όλη τη δυνατή ορατότητα στις ακροάσεις και να περιορίσουμε την μυστικότητα των συνεδριάσεων και κλεισμένων των θυρών μόνο σε, εκείνες, σε εκείνους που ζητάν εχεμήθεια. Η αρχή μας να είναι πλήρης ορατότητα για όποιον θέλει να παρακολουθήσει και να περιοριστεί πολύ ο αριθμός των μυστικών συνεδριάσεων. Μόνο όσοι το ζητάνε το ξαναλέω για να το καταλάβετε καλύτερα. Οι συντονιστές της εικόνας, λοιπόν θα το φροντίσουν. Είναι εδώ η συντονίστρια των σοσιαλιστών, μπορεί να μείνει και η βοηθός μου. Θα περιμένω άλλα πέντε λεπτά, μετά όμως θα φύγω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για αυτό το σημείο, αύριο το πρωί ξεκινάμε με τη βελγική αντιπροσωπεία στο γραφείο του Κοινοβουλίου. Bon. techniquement... Μπορούμε να βρεθούμε 8.30 ώρα αύριο το πρωί για να συμφωνήσουμε. Γιατί υπάρχει ε, τώρα μια συνεδρία στο συντονιστό ε, της ΕΚΟΝ. Και όχι μόνο η Ελίζα θα είναι απούσα, αλλά και άλλα μέλη της α, ε, αντιπροσωπείας δεν μπορούν να παραστούν. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Είτε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα ή να συμφωνήσουμε αύριο ότι θα βρεθούμε στις 8.30. Δεν μπορείτε. Έχω, με τον Υπουργό, έχω μια συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Σήμερα πρέπει να συμφωνήσουμε. Ας ξεκινήσουμε τώρα και θα ενημερώσουμε την ε, Ελίζα τηλεφωνικά. Εκτός και αν μπορείτε να μας πει αμέσως η Λίζα το πιο σημαντικό σημείο κατά την άποψή τη για τη σύσταση που πρέπει να κάνει. Για τι ε, ακροάσει μα αύριο στο Βέπιο. Δεν έχω ειδικό πρόβλημα. Αν είσαστε σε φάση να, να λάβετε αποφάσεις τώρα, Μπορείτε να μας πείτε συνοπτικά τα προβλήματά σας για να σας απαντήσω, γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις προαναγγελθήσεις επισκέψεις. Μάλιστα. Σας προτείνω λοιπόν να τελειώσει η δημόσια συνεδρίασή μας, όσοι μπορούν να μείνουν παραμένουν και αύριο το πρωί θα πω κάτι που μπορεί να το ακούσει όλος ο κόσμος. Θα συνεδριάσουμε στις 9 στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Βελγίου. Έτσι. Το γραφείο του Κοινοβουλίου στο Βέλγιο, που είναι πολύ κοντά. Από 9 με 11 θα ακούσουμε ένα πάνελ πυρογνωμόνων. Εν συνεχεία, από τις 11 και 4 θα έχουμε ένα λεωφοριάκι που θα μας πάει το επιμελητήριο, νομίζω, του Βελγίου και επί μια μισή ώρα από τις 11.30 μέχρι τη μια θα έχω μια συνεδρίαση με την Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού του Βελγικού ε, Κοινοβουλίου και συνεχεία θα μας προσκαλέσουν οι Βέλγοι Ευρωβουλευτές ε, σε ένα γεύμα για μία ώρα. Για ένα Γάλλο τώρα μία ωρίτσα για να φάει είναι λίγο σύντομο, λίγο μικρό έτσι το διάστημα που μας δίνουν. Η Ανελίζα και ο Πίτερ με κροϊδεύουν. Από τις 2 η ώρα θα πάμε να δούμε τον κύριο Στίβεν Βάνενμπερτ που είναι επικεφαλής της υπηρεσίας που ασχολείται με τα tax rulings. Από τις 2 με 3 προβλέπεται κανονικά αυτή η συνάντηση. Εγώ ήθελα, αν συμφωνούν οι να, να μείνουμε 2 ώρες με τον κύριο αυτό γιατί νομίζω ότι για το Βέλγιο, όπως και για άλλες περιπτώσεις, το πρόβλημα νούμερο ένα δεν είναι τόσο ο νόμος, αλλά ο τρόπος που εφαρμόζεται ο νόμος. Αν λοιπόν οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του, του νόμου θα μας υποδεχτούν στις 2 η ώρα στο γραφείο τους Rue de la Loi, η οδός του νόμου, έτσι, σύμβολο, σύμβολο είναι αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να του προειδοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε στι 3. Αν θα δεχθούν στι 2, αποκλεί να φύγουμε στι 3. Θα κάτσουμε πιο πολύ. Εκτό και αν ο Πίτερ έχει διαφωνία. Ένα σύντομο σχόλιο με ενημέρωσαν πως μόνο οι βουλευτές που είναι μέλη της αντιπροσωπείας μπορούν να μπουν στο επίσημο πουλμανάκι και δεν θα μπουν οι άλλοι. Θα κανονίσουμε ένα δεύτερο αμάξι λοιπόν που θα ακολουθεί το πρώτο. Από μόνοι μας. Να πω μόνο πως ποτέ δεν έχω ακούσει κάτι τόσο γελίο όσο είμαι εδώ. Έξι χρόνια δηλαδή. Εγώ είμαι 16 χρόνια εδώ, λέει ο πρόεδρος. Και έχω ε, συναντήσει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και χειρότερα. Οπότε ναι, θα το κανονίσουμε. Μάλιστα. Η δημόσια συνεδρίαση κλείνει εδώ. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια για αυτούς που θα μείνουν για την αυριανή μας οργάνωση. Ζητώ συγγνώμη, Ελίζα, που θα τα ακούσεις.